Good afternoon. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε στην κοινή αυτή ακρόαση, μάλλον το εργαστήριο, το κοινό εργαστήριο με την Επιτροπή Αναφορών και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Από κοινού θα μας απασχολήσει ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, θέματα διακρατικά σε ό,τι αφορά την υιοθεσία. Έχετε μπροστά σας το πρόγραμμα, είναι πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά πιστεύω ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακή. Η Επιτροπή Αναφορών έλαβε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών πολλές αναφορές που είχαν σχέση με διεθνείς υιοθεσίε. Ακόμα και αν ο αριθμός τους παρέμεινε σχετικά ε, χαμηλός, ε, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε, να αντιμετωπίζουμε προβλήματα που αφορούν τους πολίτες. Η Επιτροπή απάντησε ότι δεν, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρχουν διεθνείς ε, ε, κανόνες για τα θέματα αυτά από τη στιγμή που όλες οι χώρες μέλη έχουν προσυπογράψει την σύμβαση της Χάγης που λέει στο άρθρο 23 ότι μία υιοθεσία που έχει πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές ε, της χώρας υιοθεσία έχει γίνει σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης και κατά συνέπεια θα ε, τύχει αναγνώρισης ε, στο, από το άλλο κράτος. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα αλλά. Η εφαρμογή αυτής της σύμβασης είναι ένα θέμα της αρμοδιότητας της χώρας μέλους και φαίνεται ότι μερικές χώρες μέλη δεν συμμορφώνονται με αυτό. Αυτή η κατάσταση μερικές φορές οδηγεί σε παραβίαση της ελευθερίας ε, σε κυκλοφορίας και σε πρακτικά προβλήματα για τους πολίτες και για τα παιδιά που έχουν υιοθετηθεί. Αυτό λοιπόν δείχνει πόσο σημαντική είναι η συζήτηση που θα διεξαχθεί στα πλαίσια αυτού του εργαστηρίου. είναι ανάμεσά μα και ο Ταντέους Βέσκα που είναι ο αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να συμπροεδρεύσω αυτήν την συνεδρίαση, το δεύτερο τμήμα της. Όπως είπε η Σεσίλ, αυτό το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα είναι ένα από τα ουσιαστικότερα αν τα κοιτάξει κανείς ε, υπό το φως του διεθνούς δικαίου. Πρόκειται για μία από τις πιο ευάλωτες κατηγορίες πολιτών που πρέπει σήμερα ιδιαίτερα να προσέξουμε. Πρόκειται για τα παιδιά. Το θέμα της υιοθεσίας είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Αν κοιτάξει κανείς το πρόγραμμα της σημερινής συνεδρίασης, διαπιστώνει ότι οι εμπειρογνώμονες θα επεξεργαστούν θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά διαφορετικά. Θα μιλήσουμε για την διακρατική υιοθεσία, τη διεθνή υιοθεσία, αλλά και την υιοθεσία στο εσωτερικό μιας χώρας. Θα μιλήσουμε επίσης για θέματα διεθνούς υιοθεσία που αφορούν χώρες ε, μέλη της Συμφωνίας της Χάγης, αλλά και για υιοθεσία που αφορά χώρες που δεν έχουν ε, προσυπογράψει την ε, Σύμβαση του 1993. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ ευρία θεματολογία και προσωπικά πιστεύω ότι οι σημερινές μας συζητήσεις σίγουρα θα έχουν καθοριστική αξία. Σαν εισηγητής θα ξεκινήσω με τους σκιώδεις εισηγητές της ε, εργασίας μας για θέματα διεθνούς υιοθεσία. Πρόκειται για μια ιδίας πρωτοβουλία έκθεση και έχω την εντύπωση ότι η σημερινή ημέρα θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την ε, έκθεση που θα προετοιμάσω όλα αυτά τα οποία θα ακουστούν σήμερα εδώ θα συμπεριληφθούν στην έκθεση που θα προετοιμάσω. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο κανονισμός Βρυξέλλες 2 είναι σε φάση επεξεργασίας όπως και θέματα που αφορούν την ανάθεση των παιδιών, θέματα οικογενειακού δικαίου και οικογενειακού κώδικα. Οι υπάρχουσες ε, λύσεις σε διεθνές επίπεδο δεν είναι επαρκής και είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανείς ότι σε πολλούς τομείς μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε προσαρμογές έτσι ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι το ερώτημα αν θέλετε, γιατί δημιουργήθηκε το εργαλείο της υιοθεσία και εάν οι ενήλικες οι οποίοι υιοθετούν, αν θέλετε, καλύπτουν τις ανάγκες τους ε, να αποκτήσουν παιδιά. Σε κάθε περίπτωση πρωταρχική σημασίας είναι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και η βελτίωση της ε, ε, ζωής αυτών των παιδιών. Είναι δική μας ευθύνη λοιπόν να μην ξεχνάμε ποιο είναι το κύριο εγχείρημα, αν θέλετε, αυτής της νομοθεσίας, το κύριο θέμα γύρω από το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και θα ξεκινήσουμε με την κυρία Μακίνα, Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές που αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα των διακρατικών υιοθεσιών. Είναι ένα θέμα που καλούμε συχνά να αντιμετωπίσω όταν ε, καλούμε να ε, επιληφθώ θεμάτων όπως οι, όπως οι απαγωγές παιδιών. Χαίρομαι λοιπόν, μου δίνεται η δυνατότητα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Αναφορών και την Επιτροπή Νομικών ε, Υποθέσεων για την θαυμάσια συνεργασία που υπήρξε. Μιλάμε για ένα τροτό μέρος του πληθυσμού τα παιδιά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους και θα πρέπει να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δώσουμε το λόγο τώρα σε τρεις ομιλητές, την κυρία Βίσκσον, τον Μανσίσο και τον κύριο Γιάροσα. βλέπουν ε, το θέμα από εντελώς ε, διαφορετική οπτική γωνία. Θα ήθελα να στραφώ πρώτα στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, γιατί είχατε μια διερευνητική αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο και νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον για τους συναδέλφους εδώ να ακούσουν πώς πήγαν τα πράγματα και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της διερευνητικής αυτής αποστολής. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας ε, τις εμπειρίες που βιώσαμε ως Επιτροπή στο Λονδίνο. Η διερευνητική επίσκεψη οργανώθηκε πριν από μερικούς μήνες και έλαβε χώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για τις ε, δυσκολίες για να αναγνωριστεί μια υιοθεσία. Αντίθετα, θα μιλήσω για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς όταν δεν θέλουν το παιδί τους ε, να υιοθετηθεί. Θα επανέλθω όμως στο θέμα αυτό σε λίγο. Επιτρέψτε μου να σας πω πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα στην Επιτροπή Αναφορών λάβαμε περίπου 20 αναφορές που αφορούσαν περιπτώσεις παιδιών που είχαν αναλυφθεί στην Ουαλία ε, και την ε, ε, Αγγλία από ιδρύματα και που μετά δόθηκαν για υιοθεσία χωρίς τη συνένεση των βιολογικών γονιών. Γιατί ονομάσαμε λοιπόν αυτές οι υιοθεσίες μη συνενετικές ε, ή βεβιασμένες υιοθεσίες Προσπαθήσαμε πάντοτε, αυτό έγινε λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του παιδιού και αυτό είναι σημαντικό. Όταν ε, συζητάμε θέματα παιδιών θα πρέπει να έχουμε πάντοτε τη βεβαιότητα ότι δρούμε προς το συμφέρον του παιδιού. Αυτό θα πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος. Η καλύτερη λύση για το παιδί μπορεί να αλλάζει από το ένα παιδί στο άλλο. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μία εντολή υιοθεσία αυτού του τύπου είναι μη αντιστρέψιμη. Δεν υπάρχει γυρισμο σε αυτά. Φαίνεται ότι πρόσφατα παρατηρήθηκε μία αύξηση στον αριθμό περιπτώσεων ε, όπου οι γονείς δεν ήταν από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ήταν από την Ανατολική ε, Ευρώπη, Σλοβακία, ε, Λετωνία, Βουλγαρία. Και η διακρατική πτυχή καθιστά την Επιτροπή Αναφορών, αρμόδια επιτροπή για να εξετάσει αυτές τις αναφορές είναι διακρατικές, διακρατικά θέματα, όχι εθνικά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι θέματα δικής μας αρμοδιότητας. Καλέσαμε λοιπόν στην Επιτροπή μερικοί από, από όσους υπέβαλαν την αναφορά για να ε, μας ενημερώσουν και για να μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα για την κατάσταση. Ζητήσαμε από την αστυνομία να συντάξει μία έκθεση και μας υπευλήθη η έκθεση αυτή από το συντάκτη, το καθηγητή Τέμπερ από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Εγώ θα έλεγα όσοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο αυτό θέμα να διαβάσουν τη συγκεκριμένη έκθεση. Είναι μια έκθεση την οποία ε, που θεωρήθηκε ιδιαίτερα καλή όχι μόνο από εμά, αλλά και από εμπειρογνώμονες που συναντήσαμε στο ε, Λονδίνο και που έκαναν αναφορά σε αυτήν πολλές φορές. Εκτός από αυτό μια έκθεση της κοινοβουλευτική Συνέλευσης του Βουλίου της Ευρώπης δημοσιεύθηκε φέτος το Σεπτέμβριο και εκεί υπήρξε κάποιος προβληματισμός για την κατάσταση που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ιδέα λοιπόν, ε, δημιουργήθηκε έτσι η ιδέα μιας διερευνητικής αποστολής. Στόχος μας ήταν να ανταλλάξουμε απόψη με τους άμεσα ενδιαφερόμενους ή άμεσα σχετικούς για να έχουμε μια εξισορροπημένη άποψη και για να πάρουμε ε, περισσότερα στοιχεία για το κοινωνικό και νομικό σύστημα στην Ουαλία και την Αγγλία. Ε, στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν οκτώ βουλευτές. Ε, πραγματικά η αποστολή είχε οργανωθεί πάρα πολύ καλά από τη γραμματεία. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με πολλούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας τις απόψεις τους και την εμπειρία τους. Συναντήσαμε κοινωνικούς ε, ε, ε φορείς, κοινωνικές λειτουργούς, ε, αλλά και τα ε, παιδιά, προσώπους από την αστυνομία, τον ε, επικεφαλής, τον αρμόδιο για θέματα οικογενειακού δικαίου ε, εκπροσώπους των διπλωματικών υπηρεσιών της Βουλγαρίας και της Λετωνίας, εξειδικευμένους δικηγόρους στο οικογενειακό δίκαιο, δύο βουλευτές, οι οποίοι κάνουν μία εκστρατεία υπέρ των δικαιωμάτων της οικογένειας στην Ουαλία και ε, την Αγγλία. Θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα. Η πρόσβαση στα στατιστικά δεδομένα είναι δύσκολη επειδή τα δεδομένα δεν αναφέρουν, τα στοιχεία δεν αναφέρουν την εθνικότητα των γονέων. Συνεπώς δεν έχουμε μία συγκεκριμένη ιδέα του εύρους του προβλήματος όταν μιλάμε για τις δικρατικές υιοθεσίες. Κάτι που γνωρίζουμε όμω πέραν πάσης αμφιβολίας είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία μοναδική περίπτωση από τη στιγμή που το επιτρέπει να γίνουν υιοθεσίες δυστυχώς στη σύμφωνη γνώμη των γονιών. Δηλαδή η μη συνενετική υιοθεσία είναι κάτι ασύνηθες, αλλά ασύνηθες είναι και, ασύνηθες είναι και η συχνότητα με την οποία γίνεται και η ταχύτητα με την οποία γίνεται το επίπεδο των υιοθεσιών ε, στις άλλες χώρες ε, είναι πιο ε, χαμηλό και ε, χρησιμοποιείται πάρα πολύ σπάνια. Όλες οι συναντήσεις ε, που έγιναν ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, μάθαμε για το νομικό σύστημα, για τις πρακτικές των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και για τις ε, φιλανθρωπικές οργανώσεις που εμπλέκονται. Θα ήθελα όμως να σας να αναφερθώ λεπτομερέστερα σε κάτι που είπε ο Sir Μάντι πάρα πολύ γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο ως διάδοχος του Σερ Μάθιου τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αργότερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Πάρα πολλές ε, φορές ε, γίνονται αναφορές ε, στις αποφάσεις του. Δεν δίστασε να επικρίνει τις νομικές υπηρεσίες σε ό,τι αφορά θέματα υιοθεσία. Και πραγματικά είναι ένα σημείο αναφοράς για τους δικαστές οικογενειακού δικαίου θεωρεί ότι πολύ συχνά στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν κατάφεραν να ε, ε, συμμορφωθούν ε, με την σύμβαση της Βιέννης για τις προσκενικές σχέσεις και σε κάθε περίπτωση σε περιπτώσεις που δεν περιορίζονται μόνο στην Ευλόπη οι σχετικές προξενικές αρχές θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να ενημερώνονται εκτός αν η οικογένεια πει όχι η συνενέση. Εάν κάποιος ε, ξένος πρόσωπος ε, θέλει να είναι παρόν στο δικαστήριο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παρίσταται εκτός αν υπάρχουν λόγοι που υπαγορεύουν να γίνει το αντίθετο. Ο Σε Τζέιμς επίσης αναφέρθηκε στη ε, σημασία του να γίνει αναφορά στο άρθρο 15, το οποίο επιτρέπει στο Εθνικό Δικαστήριο να, μεταγράψει, να μεταφέρει τη διαδικασία σε ένα Εθνικό Δικαστήριο, ε, ε, Σύμφωνα με αυτόν, το άρθρο αυτό χρησιμοποιείται πολύ πιο συχνά στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας από ό,τι στα δικαστήρια της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ένα θέμα επί του οποίου επέμεινε και που είναι ουσιώδους σημασία σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και ιδιαίτερα σε θέματα που αυτό του οικογενειακού δικαίου είναι ο σεβασμός της πολιτιστικής διάστασης του θέματος σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις ε, δεν θέλησε να αμφισβητήσει αυτό το οικοδόμημα γιατί δεν ήταν προς το συμφέρον του παιδιού. Παρόλα αυτά ε, τον απασχολεί η προσέγγιση και των μαρτύρων και του δικαστή που θα πρέπει να είναι αυστηρό, αναλυτικό και να αναφέρεται σε τελευταία γεγονότα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η υιοθεσία επιτρέπεται ως εσχάτη λύση και μόνον αφού γίνει μία διεξοδική ανάλυση των περιστάσεων που αφορούν το παιδί, συμπεριλαμβάνοντας και θέματα που αφορούν γλωσσικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά του παιδιού ο, ο συνυπολογισμός όλων αυτών θα οδηγήσουν το δικαστήριο στο να αποφασίσει ότι αιτιολογείται μια πράξη υιοθεσία. Τέλος, ο Σερ Τζέιμς θεωρεί ότι τα πράγματα εξελίσσονται και πιστεύει ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα είναι θέματα που θα πρέπει να ανήκουν στο παρελθόν. Ή μάλλον θα ανήκουν στο παρελθόν πολύ σύντομα. Προσωπικά επιτρέψτε μου να πω ότι συμφωνώ ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει η ευημερία του παιδιού. Πιστεύω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία θα πρέπει να βοηθήσει τις οικογένειες να μείνουν ενωμένε. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να έχουν σχέση με τους γονείς τους και σχέση με την πολιτιστική και γλωσσική τους κληρονομιά στην αρχή θεωρήθηκε ότι ήταν ασυμβίβαστα όλα αυτά. Χάρη όμως αυτή την ανταλλαγή των απόψεων, τώρα η άποψή μας είναι σαφέστερη σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα και τα προβλήματα και των δύο μερών και ελπίζουμε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε κάποιες εφικτές ε, προτάσεις. Η Επιτροπή μου ε, ασχολείται με το σχέδιο έκθεσης και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σωστά εξισορροπημένο έγγραφο εργασίας το οποίο θα συνυπολογίσει τις ανάγκες όλων εκείνων που θέλουν να εξετάσουν εντελεχέστερα αυτό το θέμα. Εγώ ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ για τα ευρήματα της μελέτης σας. Είναι ενθαρρυντικό ότι όταν καλείς ε, ασχολείται και μελετά ένα θέμα, το καταλαβαίνει καλύτερα. Ελπίζω λοιπόν ότι όλα σας είναι τα μας βοηθήσει Θα ήθελα τώρα τον επόμενο ομιλητή, τον Sir Matthew Thorpe, τον οποίο, για τον οποίο, στον οποίο ήδη αναφέρθηκε η κυρία ε, να σας τον παρουσιάσω. Έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο Ηνωμένο Βασίλειο ως πρώην δικαστής ειδικό με τέτοια θέματα οικογενειακού δικαίου. Σας ευχαριστούμε Μάθιο, που είστε εδώ και θα μοιραστείτε μαζί μας την ε, πάρα πολύ πλούσια εμπειρία που έχετε και θα ακούσουμε και κάποιες από τις συστάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε. Ο τίτλος σας είναι είναι πώς θα προστατευτούν τα παιδιά και ποιες είναι οι ε, εντάσεις που δημιουργούνται πολλές φορές από την ποικιλομορφία εθνικών νομοθεσιών επί του θέματος στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι και για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση που είμαι εδώ και μου δίδεται με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να εκθέσω τις απόψεις μου σε αυτό το σεμινάριο. Όσο δικαστής επί αυτού του θέματος μπορώ να πω ότι με έχει οδηγήσει κατά τη διάρκεια όλης μου της επαγγελματικής ε, ε, καριέρας να ασχοληθώ με τέτοιου είδους ε, θέματα, πρώτα απ' όλα σε εθνικό επίπεδο, στην ε, Αγγλία και στην Ολία και μετά να είμαι διεθνής εκπρόσωπος για τέτοιου είδους θέματα. Και βεβαίως τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα τα βοήματα έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές και πρέπει να σας πω ότι πρώτα απ' όλα μία ε, γιαγιά από την Σλοβακία έκανε έκκληση ώστε να μπορέσει να υιοθετήσει το εγγονάκι Και την υπεράσπιζε στο αίτημά της αυτό η σλοβακική κυβέρνηση, την οποία, το η Σλοβακία, την οποία εκπροσωπούσε ένας δικαστής, εκπρόσωπος της κεντρικής αρμόδιας αρχής. Μία ακρόαση για ένα τέτοιου είδους θέμα πρέπει να πω ότι έχει σε συγκινησιακό επίπεδο μεγάλη επιρροή στο σύνολο των δικαστών. Υπήρχαν δύο ε, ειδικοί επί του οικογενειακού δικαίου, εγώ και ο διάδοχός μου και ένα τρίτο μέλος του δικαστηρίου και εμείς οι δύο ειδικοί επί του οικογενειακών θεμάτων είχαμε διαφορετικές απόψεις. Σε τρεις εβδομάδες συζητήσαμε το θέμα αυτό και ανθεωρήσαμε τις απόψεις μας τρεις φορές και τελικά χρειάστηκε αποφασίσουμε πριν τα Χριστούγεννα και το τρίτο μέλος του δικαστηρίου ε, ήταν με τη δική μου άποψη, τα δύο αυτά τα παιδιά, δύο ήταν τα παιδιά που έπρεπε να υιοθετηθούν, πήγαν στην ε, Σλοβακία και αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και στην μελέτη Fathom Green 3.2. Εγώ το Ιούλιο του 2013 συνταξιοδοτήθηκα και άρχισα μια νέα σταδιοδρομία ως ε, ανεξάρτητο σύμβουλο σε τέτοιου είδου θέματα. Και ήρθαν σε επαφή μαζί μου ε, για τέτοιου είδους ε, θέματα εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Πολωνίας. Στην Πολωνία επίσης είχα τέτοιου είδους επαφές για την ε, απόφαση Μέγαν. Αλλά πρέπει να σας πω ότι την ε, σφαιρική αντίληψη που έχω για το όλο θέμα και την εξέταση των δύο πλευρών την ε, απεκόμισα μετά από την υπόθεση με την οποία ασχολήθηκα για τη Σλοβακία. Στην Σλοβακία έχω διοργανώνω από κοινού μία, κάποιες ε, διασκέψεις ε, οικογενειακού δικαίου στην ε, Μπρατισλάβα, στην σχετική Επιτροπή Οικογενειακών Υποθέσεων δίνω κάποιες συμβουλές, είμαι σύμβουλος επίσης για ΜΜΕ, συνδιοργανώσα και επίσης ένα σεμινάριο το Μάιο του 2014, έφερε και πρόεδρος και επίσης και διάφορες άλλες ε, συναντήσεις ε, πριν ε, να προσχωρήσουν οι 10 νέες τελευταίες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ειδικού τέτοιου είδους θεμάτων, ε, θέματα. Επίσης, έχω ε, διοργανώσει σε επίπεδο προξενείων και Υπουργού Δικαιοσύνη, συγγνώμη, του Υπουργείου Παιδείας, διάφορα τέτοια σεμινάρια, δεδομένου ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι αυτό το οποίο εκδίδει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα που αφορούν τα παιδιά που δεν έχουν τη Βρετανική υπηκότητα αλλά είναι υπήκοοι άλλων κρατών μέλων. Επίσης έχω διευκολύνει όλες τις διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει για το ε, σύμφωνο κατανόηση Πίτερμπρο, στο οποίο θα επανέλθω. Κατά συνέπεια πρέπει να σας πω ότι έχω από τότε που έχω συνταξιδοτηθεί αποκομίσει πολλά στοιχεία και έχω μεγαλύτερη αντικειμενικότητα για τέτοιου είδους θέματα και συνειδητοποιώ ότι πρέπει να υπάρχει επικοινωνία μεγάλη και συνεργασία σε έναν τομέα τόσο σημαντικό. Η μελέτη Γκλίν δημοσιεύτηκε το 2012 και θα πρέπει να σας πω ότι ήδη έχει αποκομίσει πάρα πολύ θετικά σχόλια, δεδομένου ότι είναι διεξοδική, πλήρης και κατά την άποψή μου πάρα πολύ αξιόπιστη. Τι θα μπορούσα να προσθέσω, λοιπόν, μετά από αυτό το που έγραψε ο Δόκτωρ Φέντεν Γκλίν. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να προσθέσω είναι ε, το εξή. Οι τρει παρατηρήσει που έχω να κάνω είναι οι εξή σχέση με το θέμα αυτό. Στι 2 Νοεμβρίου έγινε μία ε, δήλωση στον τύπο εκ μέρου τη κυβέρνηση σε σχέση με το ότι οι συγγενείς ε, οι οποίοι είναι μακρινοί δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν θέματα υιοθεσία παιδιών, δεδομένου ότι πολλές ε, φορές δεν μπορούν να βρουν στις τον τρόπο αυτό τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο είπε ο υπουργό αναφορά τις προθέσεις τους. Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τους ε, εκπροσώπου του Times τότε. Στο παρελθόν, ε, το Times ήταν σαν Ευαγγέλιο για όλο τον κόσμο. And this is a quotation. Αλλά σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ελέγχθη ότι στο μέλλον όποιος συγγενής ε, προσπαθεί να υιοθετήσει ένα παιδί θα πρέπει να δείξει ότι έχει στενό συγγενικό δεσμό. Και θα πρέπει να υπάρχει ε, η απόδειξη ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν τα πάντα και να αφοσιωθούν στο παιδί που θα υιοθετήσουν. Η υιοθεσία είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό, ευαίσθητο και δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται από και να ε, γίνεται πιο δύσκολη από ε, άτομα τα οποία δεν είναι κατάλληλα ή από διά... τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη διάφορα κοινωνικά θέματα διότι δυσκολεύουν τη ζωή του παιδιού προς υιοθεσία. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μία ένταση μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας σε τέτοιου είδους θέματα και στην συγκεκριμένη αυτή εφημερίδα γίνεται κατά κάποιο τρόπο η άποψη η οποία είναι αυτή που εκφράζει και ο Πρωθυπουργό. Αυτό το οποίο λέγεται στην απόφαση Γκλίν είναι ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση με αυτό τον τρόπο λιγότερα παιδιά δόθησαν προς υιοθεσία Και η υιοθεσία θα πρέπει να είναι η ίστατη διαδικασία στην οποία καταφεύγει κανείς όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος επίλυση του προβλήματος. Και αυτό το οποίο ε, λέγει ο Πρωθυπουργό ε, ανταποκρίνεται στην ε, πολιτική της κυβέρνησης. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μία διαφορά και ένδειξη μεταξύ των δύο απόψεων μεταξύ δικαστικής και πολιτικής εξουσίας. Ο στόχος της πολιτικής εξουσίας είναι από ορθολογική πλευρά κάτι το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε. Εάν λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι πρόκειται για μία πολιτική που θα εφαρμόζεται και θα αφορά μόνο τα αγγλάκια αλλά θα πρέπει να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ μιας πολιτικής που εφαρμόζεται για τους Άγγλους υπηκόους στη συγκεκριμένη περίπτωση και των παιδιών που έχουν κάποια άλλη κοινοτική εθνικότητα. Για αυτούς χρειάζεται να έχουμε σαφείς κανόνες που θα ακολουθηθούν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο υπεύθυνο δικαστής εξέφρασε αυτή την άποψη. Τότε, από τότε που εκδόθηκε αυτή η απόφαση, έρχομαι στο δεύτερο θέμα που είναι σημαντικό. Μία on the same day as the government statement. And in και τελικά ο πρόεδρος στο τμήμα αυτό της απόφασης αναφέρει ότι σε κάποιες ε, προηγούμενες ε, υποθέσεις αναφέρεται δηλαδή στην ομολογία και αναφέρεται φυσικά στην υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τους οι εκάστοτε αποφάσεις για την τοποθέτηση ενός παιδιού σε μια οικογένεια της ε, γλώσσας, της χώρας προέλευσης και του τόπου διαμονής. Στο δικό μας σύστημα, το οποίο βεβαίως είναι τελείως διαφορετικό από τα νομικά συστήματα άλλων κρατών μελών, που βασίζονται στο αστικό δίκαιο, και ακριβώς επειδή σε μας οι δικαστές ασκούν τη διακριτική τους ευχέρεια και διατυπώνουν και την ε, ενδεχομένως δική τους άποψη για την εκτέλεση της απόφασης και ο ε, δικαστής Γκλίν αναφέρεται και στο memorandum στο οποίο σας ε, αναφέρθηκα προηγουμένως το Peterborough που φυσικά αναφέρεται στις δυνατότητες ε, ενός Δήμου, μιας κοινότητας ε, στην ε, Μεγάλη Βρετανία, στο Πίτερμπορο. Γιατί αυτή η συγκεκριμένη κοινότητα, διότι πολλοί Σλοβάκοι ζουν και εργάζονται στην κομμόπολη αυτή, μαζί με υπηκός της Λετωνίας και Πορτογάλος. Υπήρχε λοιπόν εκεί μία, αν θέλετε, κοινότητα, κυρίως από τη Σλοβακία, με τα σχολεία τους, τις υγειονομικές υπηρεσίες Θεωρήθηκε λοιπόν ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια πολύ σαφή συμβατική σχέση μεταξύ της κοινότητας αυτής και της χώρας προέλευσης της Σλοβακίας για την ε, διεκπεραίωση και την επίλυση διαφορών που αφορούσαν παιδιά από τη Σλοβακία. Αυτό βεβαίως το πρωτόκολλο, αυτό το ε, μνημόνιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν υπόδειγμα για άλλες κοινότητες. Είναι σαφής η συμβατική σχέση συνεργασίας και ουσιαστικά βοήθησε όλους τους επαγγελματίες της περιοχής του Πίτερμπορο στις σχέσεις τους με το αρμόδιο Υπουργείο. Και θα ολοκληρώσω από εκεί που ξεκίνησα. Αυτό που μπορώ να πω ότι διδάχτηκα από την ε, εργασία μου σαν ανεξάρτητος σύμβουλος είναι ότι πραγματικά χρειάζεται επικοινωνία, χρειάζεται καλύτερη κατανόηση για να υπάρξει κατανόηση των διαφορετικών νομοθεσιών, παραδόσεων και πολιτικής. Και αυτό που είναι αδιαφυσβήτητο είναι ότι όταν για πρώτη φορά η Αγγλία αντιμετώπισε δυσκολίες και προβλήματα παιδιών που έπρεπε να υπαχθούν στα συστήματα προστασίας, στην ομοθεσία ε, τη δική μας υπήρχαν πολλά δυσεπίλητα προβλήματα όπως ε, γλωσσικά, διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικές παραδόσεις, τα οποία σήμερα έχουν σε μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εντοπίζονται οι δυσκολίες και τα προβλήματα αυτά εγκαίρως Και πολλές φορές βλέπουμε ότι κοινοποιούνται πολλές υποθέσεις και σήμερα το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν το προσωπικό, οι που διαθέτουμε στις, ε, στον αριθμό των υποθέσεων που προκύπτουν και εντοπίζονται. Είχα λοιπόν ε, πολλές ε, συνομιλίες με αρμόδιους τον προηγούμενο μήνα και ρώτησα αν τα πράγματα βελτιώθηκαν, αν ε, σήμερα η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Και η απάντηση ήταν ναι, υπάρχει βελτίωση. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να σας πω είναι ότι όντως διδαχτήκαμε από τα δικά μας προβλήματα, τα ξεπεράσαμε σε μεγάλο βαθμό. Αν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με καλύτερη συνεργασία, με επικοινωνία και με διάλογο, σίγουρα θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των παιδιών και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους. Εγώ σας ευχαριστώ και νομίζω ότι η τελευταία σας φράση είναι καθοριστική για το καλό των παιδιών, όπως και αυτό που είπατε για το θέμα της επικοινωνίας. Σημαντικό γενικά στη ζωή, σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία σας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, ο κύριος Γιάρος, ο πρώην συνήγορος του παιδιού από την Πολωνία. Θα μας μιλήσει για το θέμα αυτό από την άποψη του πολωνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Ο κύριος Γιάρος είναι από το δικαστήριο της Βαρσοβίας, ε, πρώην συνήγορος του παιδιού στην Πολωνία και πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Έχετε τον λόγο κύριε Γιάρος. Ευχαριστώ. E- Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, εμπειρογνώμενες κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που διοργανώσατε αυτό το τόσο ενδιαφέρον και σημαντικό σεμινάριο, ιδιαίτερα από την άποψη των παιδιών. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας μερικές παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω την προσωπική μου άποψη, όχι μόνο ως πρώην συνήγορος του παιδιού, αλλά και ως επαγγελματίας, ο δικαστής που ασχολήθηκε με θέματα οικογενειακού δικαίου στην Πολωνία. Άκουσα τον Σερ Μάθιου το που αναφέρθηκε σε διάφορα παραδείγματα διεθνούς υιοθεσίας. Παρέθεσε το παράδειγμα της Σλοβακίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Εγώ στην επαγγελματική μου ζωή δεν ε, κλείτη να αντιμετωπίσω παρεμφερείς περιπτώσεις. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τα πράγματα, να σας τα παρουσιάσω ως δικαστής οικογενειακού ε, δικαίου και συνήγορος του παιδιού. Αυτό στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου ε, σε θέματα υιοθεσία. Θα αναφερθώ στη χώρα μου, την Πολωνία, αλλά θα κάνω αναφορά και στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Θα ήθελα σήμερα να επικεντρωθώ σε τρεις βασικές νομικές έννοιες που κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα σημαντικές και παίζουν καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς υιοθεσίες. Η πρώτη έννοια είναι η έννοια του τόπου κατοικίας του παιδιού. Σταθερή, σταθερός τόπος κατοικίας. Το δεύτερο είναι το συμφέρον του παιδιού και τρίτον το βασικό δικαίωμα που έχει το παιδί στο να ληφθεί μία απόφαση. Δηλαδή το παιδί έχει δικαίωμα να εκφέρει άποψη για όλα τα θέματα που το αφορούν. Κυρίες και κύριοι, με βάση το οικογενειακό δίκαιο, άρθρο 114, παράγραφος 2, μιλάω για το ολονικό δίκαιο, σε ό,τι αφορά την τροποποίηση, την αλλαγή της κατοικίας ενός παιδιού, η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει μόνον εάν μπορούν να δοθούν εγγυήσει στο παιδί ενός ε, οικογενειακού περιβάλλοντος. Η μεταρρύθμιση του 1995 εισήγαγε αυτό το άρθρο μετά από την υιοθέτηση από πλευράς της Πολωνίας της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού πριν από την προσχώρηση της Πολωνίας στη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1993. Στην Πολωνία η σύμβαση αυτή ετέθη σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο του 1996 με βάση το άρθρο 2, εδάφιο 2 της Σύμβασης της Χάγης ορίζεται ότι το παιδί έχει μία συγκεκριμένη μόνιμη κατοικία και αν πάει σε μία άλλη χώρα, στη χώρα υποδοχής ή στη χώρα προέλευσης των μελλοντικών γονιών του, υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει ο τόπος κατοικίας. Η σύμβαση αυτή προβλέπει ότι ότι όλα τα μέρη της σύμβασης θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτό το άρθρο. Οι χώρες όμως αυτές είναι πολλές και κατά συνέπεια είναι ε, παγκόσμια η εφαρμογή αυτού δικαίου. Σε ε, αντίθεση με το άρθρο 114 του πολωνικού δικαίου, η σύμβαση αυτή συνδέει την διεθνή υιοθεσία όχι με την αλλαγή του τόπου κατοικίας, αλλά την συνήθη κατοικία του παιδιού ή τη συνήθη διαμονή το συνήθι τόπο διαμονής του παιδιού. Αυτό είναι ένα στοιχείο ε, που έχει πολλές ε, νομικές τυχές. Στο κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει να κάνουμε αναφορά στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής, ε, στην νομοθεσία στο νόμο 2014 σε ό,τι αφορά τις ευθύνες και τις τα καθήκοντα των γονιών, ο κανονισμός αυτός αντικαθαριστά το 1344. Μιλάμε για το Βρυξέλλες 2. Η έννοια αυτή είναι σαφής ε, στην συνθήκη της Χάγης. Έχουμε την ε, σύμβαση της 1ης ε, Ιουνίου 2005 σε ό,τι αφορά τα διαζύγια. Η σύμβαση του 87 σε περιπτώσεις απαγωγής ή απομάκρυνσης του ανηλίκου είναι μια φορά στην προστασία του ανηλίκου. Και έχουμε και τη σύμβαση της 19 Οκτωβρίου του 1996 που αντικαθιστά αυτή του 61 σε ό,τι αφορά τους υπεύθυνους, τους υπεύθυνους φορείς ως προς την επιμέλεια ή την προστασία του παιδιού. Είχαμε λοιπόν, έγινε η μεταρρύθμιση του Πολωνικού Κώδικα το 2008 και εκεί ακριβώς γίνεται μνήα στον τόπο συνήθους κατοικίας. Αυτό σε ό,τι αφορά το αστικό δίκαιο και την ε, ε, ε, δικαιοδοσία σχετικά με θέματα οικογενειακού δικαίου. Το θέμα αυτό αναφέρεται και σε άλλους νόμους. Έχουμε το, το νόμο που αφορά το διεθνές δίκαιο. Παρόλα αυτά εκεί δεν ορίζεται ο τόπος κατοικίας. Ο ορισμός αυτός δεν υπάρχει. Συνεπώς αυτή η συνήθις κατοικία είναι ο τόπος όπου συγκεντρώνεται, συγκεντρώνεται οι οικογενειακές δραστηριότητες μιας οικογένειας ή ενός παιδιού. Ο τόπος συνήθους κατοικίας είναι ε, κάτι συγκεκριμένο. Έκανα αναφορά στον κανονισμό του Συμβουλίου Βρυξέλλες 2. Βρυξέλλες Α, με συγχωρείτε. Έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει μια παρέμβαση του δικαστηρίου έχουμε την απόφαση του 2009 που λέει ο τόπος συνήθους κατοικία σύμφωνα με το άρθρο 8 θα πρέπει να ερμηνευθεί ως, εκείς, ως Η συνήθις κατοικία είναι εκεί που το παιδί είναι ανσωματωμένο σε επίπεδο κοινωνικό και οικογενειακό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και θέματα διάρκειας, θα πρέπει να λάβουμε τις συνθήκες διαμονής. Όλα αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως και η εθνικότητα του παιδιού, το σχολείο, η γλώσσα καθώς και οι κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις και δεσμοί του παιδιού. Αυτό λοιπόν κρίνεται με βάση όλα ε, τα στοιχεία της περίπτωσης και κλείνει η παράθεση. Ενώπιον λοιπόν αυτής της ερμηνείας είχαμε και την απόφαση του ανώτατου ε, πολωνικού δικαστηρίου του Αρίου Πάγου σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης της Χάγης που αφορά τις περιπτώσεις απομάκρυνσης ανηλίκου η σαν ανηλίκου, γίνεται αναφορά σε αυτό το θέμα ε, στην συνήτη κατοικία λέγοντας ότι ε, είναι ο τόπος αυτός που καλύπτει τις ανάγκες του παιδιού. Η συνήθις κατοικία όμως δεν ορίζεται από την επιθυμία αυτού που φροντίζει το παιδί. Η σύμβαση της Χάγης τέτοις εφαρμογή στην Πολωνία μετά την έγκριση του άρθρου 114 οι κανόνες αυτής της ε, σύμβασης ε, υπερισχύουν των κανονοτρίτων χωρών σε ό,τι αφορά τα άρθρα του Εθνικού Κώδικα. Εάν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ αυτών των άρθρων, το Σύνταγμα είναι εκείνο που στο άρθρο 91 ρητά αναφέρει ότι η σύμβαση υπερισχύει. Σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, συνεπώς, ισχύουν οι κανόνες της ε, συνθήκης της ε, Χάγης. Η συνθήκη της Χάγης προβλέπει και την αρχή της επικουρικότητας. Η αρχή όμως αυτή είναι πολύ πιο ελαστική από ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 114 του οικογενειακού δικαίου στην Πολωνία. Υπάρχει όμως και μια πιο ελαστική ερμηνεία των δικαιωμάτων του ανηλίκου. Εδώ μιλάμε για το άρθρο 4 της σύμβασης. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι η εφαρμογή των κανόνων της σύμβασης μπορούν να, ε, μπορεί να υπάρξει μόνο όταν, αφού οι αρμόδιες αρχές των χωρών μελών ελέγξουν ότι η διεθνής λύση είναι η λύση η οποία λαμβάνει υπόψη με τον καλύτερο τρόπο το συμφέρον του παιδιού. Αυτό θα πρέπει δηλαδή να εξασφαλίζεται το, το συμφέρον του παιδιού με κάθε τρόπο. Η αρχή της επικουρικότητας της σύμβασης πως είναι διατυπωμένη με ένα πολύ πιο ελαστικό τρόπο σε περίπτωση μιας εσωτερικής υιοθεσία σε μια οικογένεια υπάρχει δυνατότητα εθνικής νομοθεσίας στην περίπτωση όμως ε, που είναι προς το συμφέρον του παιδιού η διεθνής υιοθεσία, τότε αυτή, σε αυτή θα δοθεί προτεραιότητα. Υπάρχει ένα κεντρικό όργανο στην Πολωνία που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Ε, είναι αρμόδιο το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε και τέσσερα κέντρα υιοθεσία που ασχολούνται με την εφαρμογή της συνθήκης της ε, χάγη. και τα δικαστήρια απευθύνονται σε αυτά τα κέντρα με βάση το άρθρο 4.5 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ανηλίκων. Σύμφωνα με το άρθρο 4... Οι εθνικοί φορείς θα πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε να, γίνονται, να γίνουν σεβαστές όλες οι αρχές. Σύμφωνα με το άρθρο 5 θα μπορούσε να εφαρμοστεί η συνθήκη της Χάγης μόνο αφού οι αρμόδιες αρχές διαπιστώσουν ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτή η υιοθεσία, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι το παιδί μπορεί να ταξιδέψει σε μια άλλη χώρα. Του έχει δοθεί άδεια, έγκριση να το κάνει. Έχουμε το τέταρτο κεφάλαιο της ε, συνθήκης ε, της Χάγης που αναφέρεται ιδιαίτερα στους εθνικούς φορείς που ασχολούνται με θέματα υιοθεσία. Αυτό όμως αφορά και τους ετούντες υιοθεσία. Όποιος ζητάει την υιοθεσία ενός παιδιού στο εξωτερικό θα πρέπει να αποταθεί τις αρχές της χώρας συνήθους κατοικίας του παιδιού. Σύμφωνα με τις βασικές αυτές αρχές μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι σε όλες αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψη του παιδιού. Βεβαίω, λαμβάνοντας υπόψη και την οριμότητα και την ηλικία του παιδιού. Σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό θα ήθελα να επικεντρώσω τον προβληματισμό μου που προκύπτει από τη μακρά μου εμπειρία ε, ως δικαστή. Πιστεύω ότι αυτό το δίκαιο είναι αυτό που γίνεται λιγότερο σεβαστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί η άποψή του. Λαμβάνεται υπόψη η άποψη του παιδιού με βάση την, ανάλογα με την ηλικία και την οριμότητα. Για να ληφθεί υπόψη η γνώμη του παιδιού θα πρέπει να προβλεφθεί μια ακρόαση. Αν δεν υπάρξει ακρόαση πώς θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η άποψη του παιδιού. Η άποψη του παιδιού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με βάση την ηλικία, την οριμότητα, αλλά με βάση και με βάση την κατάσταση υγείας, τη μη ενδεχόμενη αναπηρία. Όλα αυτά τα θέματα δεν θα, μπορούς δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο για τη διοργάνωση μιας ακρόασης, αφού αυτό είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Κυρίες και κύριοι, η αδικία δεν έγκυται στο γεγονός ότι γίνεται μία δίκη. Η αδικία είναι ότι όταν δεν γίνεται ε, μία δίκη, όταν δεν μπορεί να υπάρξει ακρόαση ενός ανηλίκου. Είναι λογικό να προκύψουν συγκρούσεις. Συγκρούσεις προκύπτουν όταν τα βασικά δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Μάθιου το έχει δίκιο. Ο Μάθιου Τότ είπε ότι τα πάντα εξαρτώνται από την επικοινωνία. Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε καλύτερα για να υπάρχει μια συμφωνία, για να υπάρχει ε, κατανόηση. Είναι ευσεβείς πόθη ορισμένα πράγματα. Οι χώρες που προσυπέγραψαν τη σύμβαση αυτή για τα δικαιώματα του παιδιού θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις συγκεκριμένες αρχές στο εθνικό τους δίκαιο. Γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος για τα παιδιά θα είναι καλύτερος. Ευχαριστώ. And thank Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα αυτό που είπατε ότι πρέπει να ακούμε τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι που διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη, διαφορετικά συστήματα και όντως σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει προβλέπεται η ακρόαση με τη συμμετοχή των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που είπατε και γι' αυτό και θα ήθελα καταρχήν να, να ακούσουμε όλους τους συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. θα σε ευχαριστώ που οργανώσατε αυτή τη συνεδρίαση, αυτή τη συζήτηση και σε ευχαριστώ γιατί συμμετείχα στις επισκέψεις στο Λονδίνο και όλες οι συναντήσεις που είχαμε εκεί ήταν εξαιρετικές. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί άκουσα τον κύριο Γιάρος αλλά και τον δικαστή και οι δύο παρουσιάσεις τους ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Συμφωνώ και με την διάγνωσή τους. Εδώ αναφερόμαστε σε καταστάσεις που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δικαιωμάτων του παιδιού. Και μιλάμε και για κάποιες πολύ δραματικές περιπτώσεις, ανθρώπινες τραγωδίες. Υιοθεσίε που δεν γίνονται με συνένεση, χωρίς την σύμφωνη γνώμη ούτε των γονέων, ούτε των παιδιών, χωρίς να ακουστούν τα παιδιά. Αυτού του είδους οι υιοθεσίε είναι τραγωδίες. Βλέπουμε να απομακρύνονται τα παιδιά από τις οικογένειές τους, από τα αδέρφια τους και είχα δει μια εκπομπή στην τηλεόραση στην Πολωνία που αφορούσε δύο αδέρφια οι οποίοι ξαναβρέθηκαν σε ηλικία 70 ετών. Όλη τους τη ζωή επί δεκαετίες έψαχναν ο ένας τον άλλον. Ο ένας ζούσε στην Πολωνία και ο άλλος στην Αμερική. Και ήταν τόσο συγκινητική στιγμή όταν οι δύο αυτοί αδερφοί συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας. Μία άλλη περίπτωση ήταν ε, μια γυναίκα που έψαχνε το αδερφάκι της. Όταν ήταν και οι δύο παιδιά, και τον θυμάται αμυδρά αυτόν τον μικρό αδερφό. Ο μικρός αδερφός υιοθετήθηκε χωρίς να θυμάται αν πραγματικά ε, η απόφαση ήταν απόφαση κάποιου πολωνικού δικαστηρίου. Αυτό που ξέρει είναι ότι το ψάχνει από τότε. Πρόκειται για μία περίπτωση ενός παιδιού το οποίο απομακρύνθηκε από την οικογένειά του, δεν ξέρει αν ζει, αν δεν ζει, αν βρίσκεται στην Πολωνία στο εξωτερικό. Και κοιτώντα αυτή την εκπομπή, αυτό το ντοκιμότερ σκεφτόμουν ότι πρόκειται για απάνθρωπες καταστάσεις. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη χάσει τα μέλη της οικογένειάς του στον πόλεμο, μπορεί να ξαναβρει την οικογένειά του. Αν όμως η απόφαση ενός δικαστηρίου είναι να απομακρυνθεί ένα μέλος μιας οικογένειας από την υπόλοιπη οικογένεια, είναι σχεδόν αδύνατον να ξαναβρει κανείς τα αδέρφια του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν κανείς να μπορέσει να διατηρήσει την οικογένειά του, τα αδέρφια του, πρόκειται για δώρο από το Θεό, από τη φύση, όπως θέλετε μπορείτε να το χαρακτηρίσετε, αλλά πρόκειται για δεσμούς που θα πρέπει να μην σπάνε ποτέ. Χαίρομαι που ο δικαστής Γιάρος, ειδικό σε δικαιώματα των παιδιών, είπε ότι τα παιδιά θα πρέπει να εισακόνται. Σαν δικαίωμα αυτό υπάρχει στην νομοθεσία, υπάρχει στο Σύνταγμα της Πολωνίας, αλλά βεβαίως βλέπουμε στην πράξη κάτι τέτοιο να μην υλοποιείται. Ίσως αυτό να συμβαίνει μόνο στην Πολωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στην καρδιά της υπόθεσης να είναι τα δικαιώματα των παιδιών. Τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία πραγματικά θα πρέπει να προστατεύονται με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για την σημερινή συνεδρίαση. Πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους. Και αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ενδεχομένως ε, μία σοβαρή πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες θα πρέπει να γίνουν σαφείς, θα πρέπει να είναι ανθρώπινοι και θα πρέπει να ισχύουν για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ ιδιαίτερα για την επίσκεψη που είχαμε στο Λονδίνο και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν ακούω τον ε, κύριο Θόρπ να λέει ότι στη Μεγάλη Βρετανία η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν από ό,τι φαίνεται θετικά αποτελέσματα και τα δικαιώματα του παιδιού σήμερα γίνονται σεβαστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ ε, για την ε, συμβολή σας. Ο κύριος Γιάρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου. Εγώ σαν ε, μέλος ε, της Επιτροπής Αναφορών θα ήθελα να πω ότι έχουμε πολλές αναφορές που έρχονται στην Επιτροπή που αφορούν θέματα υιοθεσίας, που αφορούν θέματα μεταφοράς παιδιών, μετακίνησής τους, αποφάσεις δικαστηρίων που πραγματικά παραμένουν χωρίς απολύτως καμία εκτέλεση, απελπισμένες οικογένειες και σίγουρα στην Επιτροπή Αναφορών βλέπουμε ξεκάθαρα την ανάγκη να δημιουργηθούν σαφείς ευρωπαϊκοί κανόνες. Έχουμε μια εσωτερική αγορά στην Ευρώπη που έχει βρει, αν θέλετε, λύσεις για την ανταλλαγή εμπορευμάτων, αγαθών. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι κάτι που το έχουμε ρυθμίσει, οι άνθρωποι μετακινούνται, μπορούν να εγκατασταθούν σε μια άλλη χώρα, να γνωρίσουν ανθρώπους, να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά. Μέχρι εκεί τα έχουμε καταφέρει. Και Εγώ δεν συμμετείχα στην επίσκεψη στο Λονδίνο, αλλά έχω κάνει παρόμοιες διερευνητικές, αν θέλετε, αποστολές και στο Βερολίνο και στη Δανία. Τα συστήματα λοιπόν είναι λίγο πολύ ικανοποιητικά. Και μέχρι τώρα είχαμε, αν θέλετε, την οτροπία ότι το κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του νομοθεσία, ρυθμίζει τις δικές τους υποθέσεις και δεν πρέπει να ανακατευόμαστε. Και δεν πρέπει και να ανακατεύουμε τα συστήματα. Η κατάσταση που μας περιγράψατε για τη Μεγάλη Βρετανία σίγουρα έδειξε ότι προβλήματα και δυσκολίες υπάρχουν και πρέπει να τα εντοπίσουμε αλλά και να τα επιλύσουμε. Ο κύριος Θόρ πολύ σωστά είπε ότι όλα εξαρτώνται από την επικοινωνία. Αυτή είναι και η δική μου εμπειρία. Και εκεί που ανησυχώ είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά να λειτουργούν με το ευρωπαϊκό σύστημα. Είναι λοιπόν πολύ θετικά αυτά τα μηνύματα, αλλά Κάθε φορά που πρόκειται για διεθνείς υποθέσεις, για διακρατικές ε, υποθέσεις, διαπιστώνουμε ότι η διαδικασία χρήζει βελτίωσης. Και μόνο έτσι μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των παιδιών. Αν λοιπόν κάτι πήγε καλά ή βελτιώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, Μ' άρεσε ιδιαίτερα αυτό που άκουσα ότι το πιο σημαντικό είναι ένα παιδί να προστατεύεται, να βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση και μόνο εάν η οικογένειά του δεν μπορεί να το ανατρέψει, να το περιθάλψει, να το προστατεύσει, μόνο σε αυτή την περίπτωση και μόνο εάν το συμφέρον του παιδιού ενδεχομένως το απαιτεί, θα πρέπει το παιδί αυτό να απομακρυνθεί από την οικογένειά του. Και μ' άρεσε πολύ και αυτό που άκουσα για την ακροαματική διαδικασία, για το πώς θα πρέπει να ακούμε τα παιδιά, αλλά και τους γονείς. Πολλές φορές διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι οι γονείς αυτοί δεν είναι σε θέση σήμερα να αναλάβουν το παιδί τους. Αλλά εάν υπάρχει, αν θέλετε, μια θετική πρόγνωση όσον αφορά την πιθανή εξέλιξη αυτής της οικογένειας, σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει η απόφαση να απομακρυνθεί το παιδί να είναι τελική και μη αναστρέψιμη. Να μπορεί δηλαδή να γίνει ανάκληση αυτής της απόφασης για υιοθεσία να είμαστε ευέλικτοι, να κοιτάμε πάντα αυτό που είπατε, το συμφέρον του παιδιού και γιατί μιλήσατε για τους πιο ε, μακρινούς συγγενείς, ε, να μην τους συμπεριλάβουμε. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι μήπως και αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να βοηθήσει το παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπατε σε σχέση με την πρακτική που ακολουθείτε από τους δικαστές. Και οι δύο αναφέρεται για την επικοινωνία που είπατε ότι διαδραματίζει στα θέματα αυτά ρόλο κλειδί. Και τι σημαίνει επικοινωνία. Συνεργασία. Και το ερώτημά μου είναι το εξή. Κατά την άποψή σας, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διεθνών θεσμικών οργάνων στον τομέα αυτό είναι επαρκής. Ή θα πρέπει σε θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας να υπάρξει πρόοδος. Και δεύτερη ερώτηση, από την ε, μεγάλη σας εμπειρία ως δικαστές, από την εμπειρία σας, ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσετε όταν έπρεπε να πάρετε αποφάσεις που αφορούν την υιοθεσία παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια αυτά και τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Σε σχέση με την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο Σεν Μάθιο, οι πολιτικές δηλαδή πρόσφατα που προσπαθούν να ε, αυξήσουν την ροή των παιδιών που δίδονται σε διάφορα ε, συστήματα υιοθεσίες. Ε, Πιστεύετε ότι αποτελούν μία καλή λύση για τα παιδιά. Για τα θέματα της εθνικότητας που αναφέρετε, δεν είμαι δεν μπόρεσα να καταλάβω εάν δύο διαφορετικές άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων παντρευτούν στη Μεγάλη Βρετανία και αποκτήσουν ένα παιδί στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει το παιδί βρετανική υπηκότητα ή έχει την υπηκότητα των ε, γονιών του. Επίσης, είπε ο, η πρόεδρος Επιτροπής Αναφορών ότι είναι μη αναστρέψιμη η οθεσία δίδεται όμως μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον ή μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο εάν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες ε, για το παιδί. Η... Κυρία Ντοργα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ίσως το ερώτησή μου έχει ε, απαντηθεί γιατί έφτασα καθυστερημένη. Συμμερίζομαι την άποψη ότι θα πρέπει να ζητείτε η άποψη του παιδιού και διαρωτώ με από την εμπειρία σας υπάρχει μια ιδεατή, μια ιδινική ηλικία από την οποία και μετά μπορούμε να ζητήσουμε την άποψη του παιδιού. Περίπου. Για ποιες ηλικίε μιλάμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέξτρομ. Ευχαριστώ. Εσείς ε, αρχίσατε την ερώτηση που ήθελα εγώ να υποβάλω. Δηλαδή, όλη η διαδικασία υιοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πάρα πολύ ε, γρήγορη αν θέλετε σε σχέση με άλλες χώρες. Κατά μέσον όρο χρειάζονται 26 εβδομάδες, πράγμα το οποίο είναι περίπου μισός χρόνος μόνο. Εάν λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε στον ε, γονιό μια δεύτερη ευκαιρία ώστε να βελτιώσει τη ζωή του για να ξαναπάρει πίσω το παιδί του, η μεγάλη πλειοψηφία μεταξύ ημών θα έλεγαν ότι επιτρέπει το σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου να γίνουν πάρα πολλές ε, υιοθεσίε ε, σύμφωνα με πάρα πολύ ε, ταχείες διαδικασίες. Όταν κάναμε την επίσκεψή μας, ήρθε ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε πολύ λίγες υιοθεσίε και η απόφαση λαμβάνεται ε, μετά από εμεινή διαδικασία. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ δύο εντελώ διστάμενες απόψεις και οπτικές γωνίες που διαμορφώνονται. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις απόψεις των άλλων εμπειρών γνώμων επί του θέματος. Επειδή υπάρχει θέμα χρόνου, θέλετε, Σερ Μάθιου, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που τέθηκαν ειδικά σε εσά. Uh, judicial communication and collaboration επικοινωνία και συνεργασία στην Ευρώπη. Θα έλεγα ότι αυτά βελτιώθηκαν θεαματικά σαν αποτέλεσμα της δημιουργίας και της διεύρυνσης του, δικτύου, διεθνούς ε, δικτύου της Χάγης. Κάθε χώρα μέλος της Ευρώπης έχει έναν δικαστή σε αυτό το δίκτυο και αυτό το σύστημα τελειοποιήθηκε και πραγματικά λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Για παράδειγμα, η Πολωνία διόρισε έναν δικαστή στο δίκτυο και αυτό ήταν πραγματικά ε, ιδιαίτερα καλό για μας γιατί έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που αφορούν πολίτες της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση που καλείται να πάρει ένας δικαστής αλλά βεβαίως ο κάθε δικαστής είναι έμπειρος και αυτό τον στηρίζει και το στηρίζει η δική του οικογενειακή ζωή και η δύναμη που παίρνει από αυτή όταν καλείται να εκδώσει πολύ δύσκολες αποφάσεις. Η πολιτική της κυβέρνησης ή μάλλον στη μελέτη Φέντογκλιν ε, αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μεγάλη ένταση από την άλλη, μεγάλη πίεση από την άλλη πλευρά θέλουμε ε, το βασικό μας μέλημα είναι το καλό του παιδιού, το συμφέρον του παιδιού και ανάλογα με την ηλικία είναι το να έχει, να μεγαλώσει ε, κοντά σε ένα ζευγάρι που αγαπάει ο ένας τον άλλον. Το θέμα είναι ότι αν η κυβέρνηση επιμείνει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά αυτό, το ζήτημα που τίθεται είναι αν αν, αν δεν συνυπολογίζονται και άλλες επιλογές που θα μπορούσαν να υπάρχουν για το παιδί και νομίζω ότι στη μελέτη Φέντογκλιν αναφέρεται αυτό το σημείο. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορά σε περίπτωση μικτή του γάμου, ας πούμε, Βρετανή μητέρα, Αγγλίδα μητέρα, Πολωνός ε, πατέρας, ας πούμε ότι διαλύεται ο γάμος. Πρακτικά δεν θα δοθεί τόσο μεγάλη σημασία στη γλώσσα ή στην καταγωγή γιατί το παιδί είναι δίγλωσσο ενδεχομένως. Τώρα, περνώντας αυτό που είπε η κυρία Wisdom, οι 26 εβδομάδες είναι αναγκαίες για να ληφθούν υπόψη ορισμένα θέματα πρόνοιας. Κατά ανάγκη εισήχθη στην έκθεση ε, Ράφτερ, γιατί το σύστημα απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο και τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν. Αν έχετε ένα παιδί εννέα μηνών και δεν ε, καταλήξετε μέσα σε ένα χρόνο, αναπτυξιακά το παιδί μετά από ένα χρόνο είναι κάτι διαφορετικό. 26 αυτές εβδομάδες είναι ένας σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν επιτυγχάνεται. Μιλάμε για μια ιδανική κατάσταση και οι διαδικασίες υιοθεσία θα έπονται των διαδικασιών που, ε, της πρόνοιας που αποτελούν ένα πρόδρομο. Ακόμα και σε περιπτώσεις ε, απαγωγής, τα παιδιά αυτά θα πρέπει να ενταχθούν σε μια πιο προσωρινή δομή στο, μέσο του, στο μέτρο του δυνατού. Προσωπικά λοιπόν πιστεύω ότι δικαιολογείται αυτός ο προβληματισμός μας του να υπάρχει μια επιτάχυνση δηλαδή ε, των ε, διαδικασιών. Βεβαίως ε, το πόσο θα κρατήσει η κάθε περίπτωση εξαρτάται από μεμονωμένους, από τον μικούς παράγοντες. Ενδεχομένως χρειάζονται έρευνες σε μια άλλη χώρα μέλος. Και ίσως αυτό θα χρειαστεί, θα, θα, σημάνει ότι θα ε, υπερβούμε το στόχο των 26 μηνών και πάντοτε ασκούνται πιέσεις ε, για πιο αργούς χρόνους σε περιπτώσεις που αφορούν παιδιά από αυτές τις χώρες μέλη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση που ένας από τους πρωταγωνιστές είναι ένα παιδί, ο στόχος των 26 εβδομάδων θα πρέπει να ειδωθεί με ένα λίγο πιο χαλαρό τρόπο και δεχομένω θα πρέπει να αφαιθεί μεγαλύτερο περιθώριο για αξιολόγηση. Δηλαδή στην ουσία συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιάρης. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους παρεμβαίνοντες για τις τόσο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τους. Για να απαντήσω θα ήθελα κυρίως να βασιστώ σε ένα διεθνές κείμενο που έχουμε, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, που βασίζεται βασικά σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, στην προστασία του και την πρόσφυση των δικαιωμάτων του και η δεύτερη αρχή είναι το γεγονός ότι πρέπει να βοηθηθεί η οικογένεια από το κράτος. Η οικογένεια είναι η φυσική αιστεία στην οποία αναπτύσσεται ένα παιδί. Και μιλώ με μεγάλη περηφάνεια για το έγγραφο αυτό, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο μέρος σε πρωτοβουλία Πολωνών και κυρίως ε, του φημισμένου Πολωνού παιδαγωγού Μουρτσάφσκι, ο οποίος βρίσκεται στη φιλοσοφική βάση, αν θέλετε, του κειμένου αυτού. Η συνεργασία που αναφέρθηκε, δηλαδή είναι επαρκή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι επαρκής. Παρά το γεγονός ότι έχει επικυρωθεί από σχεδόν όλα τα κράτη του κόσμου η σύμβαση αυτή, πρέπει να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν κάποια κράτη που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού, την υιοθεσία, άλλα θέματα παρουσίας του παιδιού στα δικαστήρια, διότι το θέμα της ερμηνείας της οικογένειας είναι κάτι διαφορετικό ίσως για κάποιους. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα ώστε το, η σύμβαση αυτή να μην αντικαταστήσει τα συστήματα κοινωνικής προστασίας των παιδιών. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δούμε περιπτώσεις οι οποίες για οικονομικούς λόγους κάποιο παιδί κάποια οικογένεια χάνει το δικαίωμά της να έχει παιδί. Το παιδί λοιπόν το εμπιστεύονται σε κάποιον άλλο. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι απαράδεκτο. Αντιθέτως το κάθε κράτος θα πρέπει να βρει τρόπους να βοηθήσει την οικογένεια. Και το λέγω αυτό και από την δική μου πρακτική εμπειρία. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που επειδή ήταν πάρα πολύ φτωχή η οικογένειά τους χρειάστηκε να τα αποχωριστούν. Νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι οικονομικές συνθήκες στις οποίες ζει η οικογένεια. Δεν ξέρω, ο πρόεδρος κοινότητας, ο δήμαρχος της μικρής πόλης στην οποία ζει μια οικογένεια θα πρέπει να βοηθήσει την οικογένεια να βελτιώσει την καθημερινότητά της, να τη βοηθήσει να αποκτήσει μπάνιο. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Βεβαίως, νομίζω ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού και να οργανώνουμε και να πηγαίνουμε σε διασκέψεις διεθνείς που οργανώνονται ώστε να μάθουμε να προσπιζόμαστε καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών. Επίσης υπάρχει ένα άλλο δικαίωμα το οποίο δεν αναφέρουμε πολύ το δικαίωμα της ταυτότητας του παιδιού. Δηλαδή, σε περίπτωση υιοθεσία. Μπορεί να πει κάποιος ότι κάποιο παιδί δεν έχει το δικαίωμα να γνωρίσει την, τον τόπο καταγωγής του ή τους βιολογικούς του γονείς. Διαπιστώσαμε όμως με και είπαμε ότι τουλάχιστον στην Πολωνία εμείς δεν θα καταστρέφουμε τα, ε, τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως φερρυπίν του παιδιού, τα οποία διατηρούνται από το σχετικό οργανισμό και μετά από την ενηλικίωσή του το παιδί έχει το δικαίωμα να τα συμβουλευτεί. Δεν μπορεί κανείς να αποκόψει έναν άνθρωπο από τις ρίζες του. Νομίζω ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να το σκεφτούν το θέμα αυτό. Ίσως αυτή η πολωνική λύση να είναι μια καλή λύση. Θα μπορούσαμε όμως να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να βρούμε άλλες παρεμφερείς ακόμη και καλύτερες λύσεις. Επανέρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα. Από ποια ηλικία μπορεί κανείς να ζητήσει την ε, άποψη του παιδιού. Θα σας απαντήσω με απόλυτη σαφήνεια. Οποιαδήποτε παιδί θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ακουστεί ακόμη και τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να εκφράσουν πλήρως την άποψή τους, κυρίως αυτά τα παιδιά. Ένα παιδί, Φερρυπίν, το οποίο έχει μία κάποια αναπηρία, δεν θα το ακούσουμε επειδή έχει δυσκολίες ε, έκφρασης. Το οποίο παιδί αυτό θα πρέπει όλος ιδιαίτερος να σκεφτούμε πώς θα το προστατέψουμε και να το προστατεύσουμε. Σήμερα νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν προσυπογράψει τη σύμβαση του παιδιού πιστεύουν ότι θα πρέπει το παιδί, στο παιδί να δώσουμε όλες τις δυνατότητες να εκφραστεί. Διότι υπάρχει η γλώσσα του σώματος, η γλώσσα της έκφρασης των ματιών. Τώρα, ε, αν λαμβάνεται υπόψη αυτό που θέλει να εκφράσει το παιδί είναι ένα άλλο θέμα. Τελειώνω κυρία Πρόεδρε. Ένα παιδί 13 ετών έχει την ε, άποψή του και μπορεί να πει εάν ναι ή όχι συμφωνεί με την υιοθεσία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Δίξτον, τον κύριο Γιάρος, τον σε Μάθιου Θόρπ. Εάν μπορώ να συνοψίσω κάποια από τα σημεία αυτά σε ένα λεπτό, θα έλεγα ότι... Σε γενικές γραμμές, η εμπειρίες και η ιστορία των κρατών μελών διαφέρει. Πολλές φορές ε, υπάρχουν δυσκολίες που ουσιαστικά προέρχονται <clears throat> από το παρελθόν. Πριν από 30-40 χρόνια συνέβησαν κάποια πράγματα τα οποία ε, κάποιοι σήμερα θα πρέπει να γνωρίζουν για να τα αποφύγουν. Η κατάσταση, ακούσαμε, στη Μεγάλη Βρετανία βελτιώνεται. Στο επίκεντρο των προσπαθειών μας πρέπει να βρίσκεται το παιδί. Το παιδί και το συμφέρον του, τα δικαιώματά του. Κύριε Γιάρος, είπατε επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απομακρύνονται τα παιδιά για οικονομικούς λόγους από τις οικογένειές τους. Και πολλές φορές αυτό γίνεται χωρίς βεβαίως αυτό να είναι ο σκοπός των κοινωνικών υπηρεσιών. Επειδή και όλοι εμείς, εκτός από πολιτικοί, είμαστε και άνθρωποι και επειδή τελικά θέλουμε να συνεισφέρουμε στην εξέβρεση λύσεων, από τη μία αναγνωρίζουμε την επικουρικότητα και τις διαφορετικές παραδόσεις και ε, ευαισθησίες, θα πρέπει παρόλα αυτά να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τις επιμέρους αυτές οι υποθέσεις να βρουν μια ικανοποιητική σε ευρωπαϊκό επίπεδο της. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μαγκίνας, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό και διαπιστώσαμε ότι το θέμα αυτό προκαλεί πάθος, συγκίνηση και περνάμε στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας που είναι αυτές οι διακρατικές υιοθεσίες. Ένα θέμα που σαφώς συμπεριλαμβάνει πολλές πτυχές που αφορούν την οικογένεια. Θα επικεντρωθούμε εδώ στο θέμα του ορισμού της οικογένειας που διαφέρει στις χώρες μέλη στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οικογενειών και θα δώσω αμέσως το λόγο στον Τζιάν Πάολο Ρωμάνο από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, ο οποίος θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υποδέχεται έναν καθηγητή από Ελβετικό Πανεπιστήμιο. Έχω και Ιταλική εθνικότητα και με ευχαρίστηση είμαι εδώ για να υπηρετήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Σελήν Σατό, η οποία προσκάλεσε για να την ευχαριστήσω για τη βοηθειά της. Μου ζητήσατε να ε, παρέμβω για την ε, αναγνώριση κάποιων ε, οικογενειακών καταστάσεων. Είναι πολυσχεδής όρος κατάσταση, γι' αυτό εγώ προτιμώ τον όρο οικογενειακή κατάσταση που είναι κάτι που αφορά δύο άτομα τα οποία έχουν ε, κάποια σχέση μεταξύ τους η οποία έχει θεσπιστεί από κάποια διοικητική ή δικαστική αρχή. Σκέφτεται κανείς το γάμο ή τη συμβίωση ε, είναι η κατάσταση την οποία μπορού, στην οποία μπορεί κανείς να καταλήξει σε περίπτωση ε, διαζυγίου ή άρνησης ε, πατρότητας. Το θέμα της υιοθεσία αφορά επίσης ένα διπλό θέμα, δεδομένου ότι καταργεί ένα προηγούμενο δικαίωμα και δημιουργεί ένα νέο δικαίωμα, και ε, έχουμε περιπτώσεις, σε τέτοια περίπτωση που αφαιρείται η νόμιμη ε, ιδιότητα η γονική στους βιολογικούς γονείς και εκχωρείται στους γονείς που υιοθετούν. Θα ήθελα να ε, πω ότι υπάρχουν διάφορες νομικές επιπτώσεις από τέτοιου είδους κατάσταση. Σήμερα δεν ε, υπάρχει ένα ευρωπαϊκό νομικό μέσο το οποίο αφορά την ε, διεθνή αρμοδιότητα που μπορεί να δοθεί σε τέτοιου είδους ε, περιπτώσεις διαφορετικών οικογενειακών καταστάσεων. Δεν υπάρχουν κοινέ διατάξεις λοιπόν όσον αφορά την αναγνώριση των γάμων και των συμβιώσεων οι οποίες, ή της νομικής αναγνώρισης της υιοθεσίας ή της αναγνώρισης της πατρότητας. Υπάρχουν δύο κανονισμοί που αναγνωρίζουν την, ε, το γεγονός ότι μία κατάσταση πάβει να υφίσταται ε, όταν υπάρξει ακύρωση του γάμου ή διαζύγιο. Ο κανονισμός Βρυξέλλες 2 έχει σχέση με την αναγνώριση σε τέτοιου είδους θέματα και αφορά το, δικαίωμα, το, δίκαιο το οποίο ισχύει σε περίπτωση ε, διαζυγίου και θεσπίζει τις κανόνες οι οποίοι είναι σε ισχύ σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εκτός από τον κανονισμό Βρυξέλλες 2 υπάρχει και η σύμβαση της Χάγης η οποία αφορά τέτοιου είδους θέματα. Για να συνοψίσω, σήμερα ένα κράτος μέλος ετήσει ενό από τα δύο ενδιαφερόμενα μέλη και των δύο είναι ελεύθερο να αποφασίσει, να του χορηγήσει μια ειδική οικογενειακή κατάσταση, ενώ ένα άλλο μέρος είναι ελεύθερο να μην την αναγνωρίσει. Πολλές φορές υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες πραγματικά θεωρούνται ως καταστάσεις που χωλένουν και οι λύσεις που, που ακολουθούνται και αυτές χωλαίνουν. Θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα. Την κατάσταση του κυρίου Ντουπάν, Γάλλου και του κυρίου Μπιάνκη, Ιταλού. Σήμερα είναι ελεύθερο κανείς ε, στη Γαλλία να συνάψει ε, γάμο ε, μεταξύ ομοφύλων. Έτσι, ο Ντυπών και ο Μπιάνκι παντρεύονται στη Γαλλία, αλλά η Ιταλία για λόγους εθνικής τάξης δεν το αναγνωρίζει αυτό. Άρα, στο ε, ληξιαρχείο οικογενικής κατάστασης του κυρίου Μπιάνκι δεν αναγνωρίζει ως σύζυγό του τον κύριο Ντυπών. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι επιπτώσεις από αυτή τη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση αυτών των δύο ατόμων που είναι παντρεμένοι για την Ιταλία και σε ελεύθερη συμβίωση για την Ιταλία. Για την Ιταλία. Ο κύριος Μπιάνκι δεν έχει την υποχρέωση να δώσει διατροφή στον κύριο Ντυπον εάν χωρίσουν. Αντιθέτως, για την Γαλλία, ο κύριος Μπιάνκι είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Αν ο κύριος Ντυπον σύμφωνα με μία απόφαση της Γαλλίας. Ε, μπορεί να ζητήσει διατροφή από τον κύριο Μπιάνκι, εκείνος αντιθέτως μπορεί να ζητήσει από ε, τα δικαστήρια στην Ιταλία να ε, μην αναγνωρίσει αυτή την απόφαση. Για ποιο λόγο. Διότι εάν η δημόσια τάξη στην Ιταλία είναι αντίθετη προς την αναγνώριση αυτού του γαλλικού γάμου, μπορεί επίσης να αρνηθεί να αναγνωρίσει και το δικαίωμα διατροφής. Έτσι, αυτή η διαμάχη μεταξύ των δύο κρατών θα δημιουργήσει μία διαμάχη όσον αφορά την απόφαση που αφορά την διατροφή. Και τη στιγμή την οποία μιλούμε εμείς δεν υπάρχει κανένα νομικό μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να αποφανθούμε σε τέτοιου είδους προβλήματα μεταξύ δύο κρατών μελών. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητα. Έτσι λοιπόν... Ε, ο κύριος Ντυπών και ο κύριος Μπιάνκι δεν ξέρουν απολύτως ούτε ποια είναι όλα τα δικαιώματά τους, ούτε όλες τις υποχρεώσεις. Κάποια στιγμή ελπίζουμε ότι τέτοιου είδους πόλεμος, αν υπάρχει, θα σταματήσει. Αλλά η απόφαση ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει απαραίτητο να είναι νομική. Ίσως ε, τότε ο νόμος του πιο ισχυρού και του πιο πονηρού και του πιο ταχαίως ε, θα επικρατήσει και τότε ο κύριος Μπιάνκι για να μπορέσει να μην εκτελέσει τη γαλλική απόφαση θα μεταφέρει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία στην Ιταλία. Τώρα, εάν πεθάνει ο κύριος Μπιάνκι για τη Γαλλία ο κύριος Ντυπών, ο σύζυγος του κυρίου Μπιάνκι είναι ο νόμιμος κλειονόμος του. Για τη Γαλλία, την Ιταλία όμως του ο αδερφός του και οι αδερφές του και οι αδελφοί του είναι εκ των πραγμάτων και οι κληρονόμοι του. Για την Ιταλία δεν είναι σύζυγος του κυρίου Μπιάνκι ο κύριος Διπών. Ας υποθέσουμε τελικά ότι ο κύριος Διπών και ο κύριος Μπιάνκι υιοθέτησαν ένα μικρό Σενεγαλέζο στη Γαλλία που είναι βιολογικό ε, παιδί της κυρίας Μπέγκ που καταρχάς ε, έδωσε το παιδί της ε, για υιοθεσία, αλλά μετά το μετάνιωσε. Ο, αν πεθάνει ο κύριος Μπιάνκι υπάρχει μια, πρόβλημα όσον αφορά την κυδαιμονία του παιδιού μεταξύ της κυρίας Μπέν και του κυρίου Ντυπών. Από την άποψη της Γαλλίας που ε, αποφάσισε για την υιοθεσία και ε, την εξέδωσε τη σχετική απόδοση, ο κύριος Ντυπών είναι ο νόμιμος γονιός. Από ιταλικής πλευράς η κυρία Μπέγκ είναι η νόμιμη μητέρα. Διότι η αγκαλική υιοθεσία δεν έχει καμία αξία στην Ιταλία. Τέτοιου είδους ε, καταστάσεις συμβαίνουν και ε, νομίζω ότι είναι αντίθετες με τον στόχο μας να μπορέσουμε να έχουμε στην Ευρώπη ένα χώρο δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας. Νομίζω ότι έτσι ε, αρνούμεθα σε κάποια άτομα να βρουν λύσεις στο πρόβλημά τους, δεδομένου ότι υπάρχει θέμα ε, διαφοράς ε, διευρωπαϊκής. Είμαστε ενωμένοι στην ποικιλομορφία είναι το σλόγγαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως συγκεκριμένη περίπτωση η Γαλλία και η Ιταλία δεν είναι ενωμένε παρά την ποικιλομορφία τους, δεδομένου ότι έχουν μια διαφορετική αντίληψη περί γάμου βρίσκονται σε διαμάχη. Έτσι λοιπόν έχουμε μία διαμάχη μεταξύ νομικών τάξεων. Και εδώ έχουμε την, ε, ένα μεγάλο πρόβλημα στο δίκαιο. Πρόκειται για υποχώρηση του δικαίου. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις για να μπορέσω να βελτιώσω την ευρωπαϊκή οικογενειακή κατάσταση που αφορά τους πολίτες και αυτούς που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες από τις προτάσεις μου πάρα πολύ σύντομα. Σύμφωνα με μια πρώτη προσέγγιση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συνεχίζει να επιτρέπει σε ένα κράτο μέλος να δημιουργήσει αυτή την έννοια της οικογενειακής κατάστασης, αλλά θα πρέπει να επιτρέψει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να μην την αναγνωρίζει. Ε, θα έπρεπε η, Ευρω... η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να επιτρέψει στον καθένα να ακολουθήσει το δικό της ε, ισχύον καθεστώς. Σε αυτή την περίπτωση η Γαλλία θα πρέπει να συνεχίσει να αναγνωρίζει το γάμο του κυρίου Ντυπών και του κυρίου Μπιάνκι, αλλά η Ιταλία να συνεχίσει να αρνείται να την αναγνωρίσει. Στάτη quo λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Εάν ο νόμος που εφαρμόζεται για την, ε, διατροφή, την, υποχρέωση διατροφής ακολουθεί την γαλλική νομοθεσία, η, η Ιταλία θα έπρεπε να αναγνωρίσει ε, σε αυτή την περίπτωση τον γάμο μεταξύ των δύο ατόμων. Εάν ε, δεν μπορέσει όμως η η Ιταλία να εφαρμόσει, να εκτελέσει μία γαλλική απόφαση και να υποχρεώσει τον κύριο Μπιάνκι να δώσει την διατροφή, ε, με μια κατάσταση μεταβλητής γεωμετρίας όπως λέμε, δηλαδή μια μεσοβέζικη κατάσταση. Για, κάποιους, ε, για κάποια θέματα, σε αυτή την περίπτωση ο κύριος Ντυπών και ο κύριο Μπιάνκι είναι σύζυγοι, στην Ιταλία όπως και στην Γαλλία, αλλά για άλλα θέματα δεν θεωρούνται σύζυγοι, ούτε στην Γαλλία ούτε στην Ιταλία. Δεύτερη πρόταση. Ε, έχουμε μία περίπτωση υιοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δύο μητέρες ε, που θέλουν να υιοθετήσουν είναι μία Βουλγάρα και μία Πολωνέζα που ζουν στην Αγγλία. Εδώ το δίκαιο που ισχύει είναι το δίκαιο της Βουλγαρίας και της Πολωνίας και κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι αντίθετο αυτό προς τη δημόσια τάξη. Τώρα, αν μια Γερμανίδα θέλει να βρει μια παρένθετη μητέρα στην Ελλάδα και μπορούν οι ελληνικές αρχές να το επιτρέψουν, η απόφαση της Ελλάδας πρέπει να εκτελεστεί και και τις γερμανικές αρχές. Εάν κάτι τέτοιο γίνει θα έχουμε να κάνουμε μια σημαντική καινοτομία. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή μια τέτοιου καινοτομία θα πρέπει κατά την άποψή μου να αποδείξει ποιες είναι οι σχέσεις που απαιτούνται να υπάρχουν μεταξύ των ατόμων που θέλουν να ε, προχωρήσουν σε μια τέτοιου είδους πράξη. Αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει ώστε να αποθαρρυθεί ο τουρισμός για να βρει κάποιο σύζυγο να παντρευτεί, για να υιοθετήσει ή για να μπορέσει να αποκτήσει ένα παιδί. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν σαφείς κανόνες ώστε να έχουμε μια κατάσταση που θα γίνει όλο και περισσότερο πιο ομαλή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε για, τις, ε, για τους γάμους ε, τους, ε, μεταξύ ετεροφύλων που αναγνωρίζονται παντού ή για την ε, ε, η υιοθεσία μεταξύ συζύγων να ακολουθήσει έναν νέο κανόνα βάσει του οποίου θα λάβει την απόφασή της ή την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής ενός από τους ενδιαφερομένους για τους γάμους ομοφύλων ή για την υιοθεσία από ένα ζευγάρι ομοφύλων θα πρέπει να υπάρχει με μια διπλός κανόνες που να ακολουθείτε από την χώρα που είναι πιο ανεκτική. Τώρα, μία ε, τρίτη απόφαση αφορά τι ακριβώς θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση αυτή που σας ανέφερα που μια Γερμανίδα έχει, θέλει να βρει μια παρένθετη μητέρα στην Ελλάδα. Πριν να γίνει κάτι τέτοιο, οι ελληνικές αρχές θα έπρεπε να έρθουν σε επαφή με τις γερμανικές αρχές ώστε να δουν αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους. Αλλά αν υπάρχει διαφωνία, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Τέταρτη ε, εναλλακτική λύση, να ακολουθήσει κανείς το δίκαιο το οποίο τον ε, εναλλακτικό δίκαιο, αν μου επιτρέψετε να το ονομάσω έτσι, το οποίο θα μπορούσε να ακολουθηθεί ε, χωρίς να μπορεί βεβαίως να αντικαθιστά τα δίκαια στα κράτη-μέλη. Αυτό το εναλλακτικό δίκαιο θα μπορούσε ή θα έπρεπε να συνοδεύεται από τη δημιουργία ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες θα πρέπει να χειρίζονται τέτοιου είδους θέματα με τη βοήθεια ειδικών σε θέματα ε, μητρών καταγραφής οικογενειακής κατάστασης ώστε να μπορεί να γίνεται ένας ευρωπαϊκός γάμος, ευρωπαϊκά δικαστήρια που να ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα όπως υιοθεσίες και να υπάρχει ένα τέτοιο ειδικό καθεστώς που να αφορά και ειδικά δικαστήρια τα οποία θα ασχολούνται τέτοιου είδους θέματα. Ε, θα πρέπει τότε να υπάρχει απόλυτη αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των δικαστή αποφάσεων αυτών των δικαστηρίων. Θα πρέπει να υπάρχει μια κεντρική διοίκηση στο Παρίσι και δύο τμήματα στο Λονδίνο και στο Μόναχο. Και περιφερειακές διοικήσει στο Χόλμη για τον Βορρά και σε μια χώρα του Νότου για τον ε, ε, Νότο. Επίσης, πρέπει να πω ότι για να εφαρμόσουμε τέτοιου είδους θέματα στο οικογενειακό δίκαιο, θα πρέπει να διανύσουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο και να δούμε κατσόν δεν θα πρέπει... να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο για να δούμε πώς θα βρούμε λύσεις από τότε που υπεγράφει η συνθήκη του Άμστερνταμ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για την διαθέτηση διακρατικών θεμάτων, πράγματα οποία μας φαίνονταν αδύνατα πριν από 20 χρόνια. Ίσως και σε αυτό το τομέα λοιπόν θα μπορούσαμε να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ γιατί μας δίνεται μια διαφορετική οπτική γωνία σε αυτό το πρόβλημα. Εγώ μπορώ να προσθέσω απλώς ότι όλα όσα παρουσιάσατε βεβαίως μπορεί να αφορούν και άλλες χώρες εκτός από τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εναρμονίσουμε την ομοθεσία των κρατών μελών στον τομέα αυτό και βεβαίως <coughs> δεν πρόκειται για καθαρή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα όταν αναφερθήκατε στον κανονισμό, σκοπός είναι να δοθούν στα δύο μέρη οι δυνατότητες προστασίας και όχι να επικρατήσει ο πιο ισχυρός σε μια περίπτωση διαζυγίου, παραδείγματο χάρη, η επιλογή του δικαστηρίου και του τόπου αρμοδιότητα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλέγεται βάσει άλλων αντικειμενικών κριτηρίων. Αλλά και στον κανονισμό Ρώμη 3, αλλά και στην σύγκριση που κάνατε με τα διπλώματα τεχνίας, ουσιαστικά πρόκειται για τη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασίας Και βεβαίως ε, κανείς δεν μας απαγορεύει εδώ να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε. Θα ακούσουμε την κυρία Λάουρα Μαρτίνες Μόρα, η οποία είναι στην ε, μόνιμη αντιπροσωπεία για την σύμβαση της Χάγης. Πρόκειται για τα δικαιώματα των παιδιών σε περιπτώσεις διεθνούς υιοθεσία και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε και κάποιες νέες λύσεις που ενδεχομένως μπορεί να είναι αποτελεσματικές. Ας δούμε λοιπόν πώς έχει η σύμβαση. Θα μιλήσω στα ισπανικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό για μένα που βρίσκουμε εδώ μεταξύ εμπειρογνωμόνων εξ ονόματος της, ε, της διάσκεψης της Χάγης και αναφερόμενη στην διεθνή συνεργασία μεταξύ της δικής μας του δικού μας οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μιλήσω καταρχήν για τους στόχους, την εφαρμογή και τα συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης της Χάγης. Κατόπιν θα αναφερθώ στην αυτόματη αναγνώριση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Τρίτον, θα σας παρουσιάσω κάποιες ιδέες και σκέψεις για το μέλλον. Ο δικαστής Γιάρος παρουσίασε το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης και δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε. Θα ήθελα μόνο να σας πω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ο συνήθις τόπος διαμονής, όχι μόνο του παιδιού αλλά και των ε, υποψήφιων γονέων. Δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί κριτήριο η ηθαγένεια, αν πρόκειται δηλαδή για γονείς ε, και παιδί ίδιας ηθαγένειας. Εγώ παραδείγματος χάρη είμαι Ισπανίδα, ο σύζυγός μου είναι Ιταλός και ζούμε στην κατοχώρα. Εάν θέλω να υιοθετήσω ένα παιδί από τη Λιθουανία, αρμόδια είναι η χώρα συνήθως διαμονής. Η Ολλανδία δηλαδή. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις αρχές της Ιταλίας και της Ισπανίας για να δούμε τι θα συμβεί με την ηθαγένεια του παιδιού καθότι δεν ρυθμίζεται από τη Σύμβαση της Χάγης το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες ε, πρακτικές και εάν βρεθούμε αντιμέτωποι με διεθνείς υιοθεσίες, όλες οι εμπλεκόμενες χώρες θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαδικασία. Αυτό που κάθε φορά προσπαθώ να πω είναι ότι η Σύμβαση της Χάγης συμπεριλαμβάνει διάφορα κεφάλαια όμως είναι πάρα πολύ σημαντική η ημερομηνία του 1993. Πρόκειται για την προστασία των παιδιών. Πρόκειται για μια σύμβαση για την προστασία των παιδιών και ήδη αναφερθήκαμε στην σημασία της προστασίας των παιδιών. Το δεύτερο τμήμα αφορά την συνεργασία. Δηλαδή θέλουμε τα κράτη να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να μιλούν μεταξύ τους ώστε να αποφεύγουν τα προβλήματα. Τι κάνει αυτή η σύμβαση. Θεσπίζει ελάχιστες εγγύησεις για την υιοθεσία των παιδιών. Παναφέρθηκαν πάρα πολλά παραδείγματα στο πρώτο μέρο. Πρώτα απ' όλα η... το ότι συνενούν οι αρχές ή η βιολογική οικογένεια. Πρέπει να είναι ελεύθερη συνένεση. Ε, χωρίς να υπάρχει κανένα αντάλλαγμα, να γίνεται γραπτός και να, αφού έχει ενημερωθεί πλήρως ο Θένας. Επίσης, είπαμε ότι θα πρέπει όλες οι πληροφορίες που αφορούν την υιοθεσία να φυλάσσονται, διότι είναι πολύ σημαντικό όταν το υιοθετημένο άτομο θέλει να έχει πληροφορίες για την υιοθεσία του, να του δίνουμε απάντηση. Επίσης, μιλήσαμε για την αρχή της επικουρικότητας της διεθνούς υιοθεσίας και πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, ακούσαμε να, πόσο σημαντικό είναι να ακούγεται το παιδί ή να το επιτρέπουμε για την υιοθεσία να εκφράσει την άποψή του. Αυτό το οποίο κάνει η σύμβαση αυτή λοιπόν είναι να θεσπίζει ελάχιστες εγγύησεις, βασικές εγγύησεις. Φερρυπίν, η μητέρα μπορεί να συνενέσει στην υιοθεσία μόνο μετά από την γέννηση του παιδιού. Δεν λέγεται πότε, μετά από ένα λεπτό, μετά από δέκα μέρες, δύο μήνες. Κάθε χώρα το διαθετεί αυτό το θέμα. Η συνθήκη αυτή της Χάγης είναι πάρα πολύ ευέλικτη αν θέλετε, διότι επιτρέπει σε κάθε χώρα να ρυθμίζει κάποια θέματα σχετικά σε σχέση με την νομοθεσία του. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερος στόχος. Να αποφεύγονται καταστάσεις όπως διακίνηση ε, παράνομη των παιδιών. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχει το χρήμα. Και όταν υπάρχει χρήμα στη μέση πάντα υπάρχουν προβλήματα. Τρίτος αντικειμενικός στόχος. Να υπάρξουν επίσημοι διάβλοι συνεργασία. Να ξέρουμε με ποιον μιλούμε. ποιο είναι ο συνομιλητή μα στην άλλη χώρα. Να ξέρουμε σε ποιον θα ζητήσουμε την απάντηση σε ερωτήσει που έχουμε. Εάν όλε αυτέ οι εγγυήσει λοιπόν γίνουν σεβαστέ, σε, θα μπορούμε και μόνον τότε θα μπορούμε να έχουμε την αυτόματη αναγνώριση. Αυτόματη αναγνώριση που δίδεται στις 95 χώρες που έχουν προσυπογράψει τη σύμβαση. Φτάνουμε τις 100 χώρες. Ελπίζουμε ότι θα γίνουν 96 σε λίγες μέρες αυτές οι χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχουμε τρεις χώρες όπως η Ρωσία, το Νεπάλ και η Κορέα που υπέγραψαν αλλά ακόμη δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση αυτή. 95 είναι ένα σημαντικός αριθμό χωρών. Πολύ σημαντικός διότι όλε οι χώρες υποδοχής είναι μέλη που έχουν προσυπογράψει. Επίση είναι σημαντικό να πούμε ότι η Αφρική που, που είναι σαν τα νέα σύνορα της διεθνούς υιοθεσίας, διότι βλέπουμε ότι οι χώρες ώρες ώρες βάζουν όρια και θέλουν να κάνουν αυτό το οποίο γίνεται αυτή την στιγμή στην Αγγλία. Θέλουν κάθε παιδί να μένει με την οικογένειά του. Κάνουν όλη αυτή την δουλειά και βλέπουμε ότι πολλές φορές μπορούν οι χώρες να δώσουν μια διεθνή απάντηση στο ερώτημα και να μην μπορούν τα παιδιά να δοθούν ε, στο εξωτερικό για υιοθεσία. Και πολλές χώρες ξέρουμε ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να υιοθετήσουν παιδιά. Η Αφρική ξέρει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή έχουμε 16 χώρες από την Αφρικανική Ήπειρο που είναι χώρες που έχουν αποφασίσει να προσχωρήσουν σε σύμβαση αυτή. Υπάρχουν πολλές άλλες ε, χώρες, όπως θα εξηγηθεί αργότερα, που δεν ε, προβλέπουν την υιοθεσία, άρα δεν είναι μέλη. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Βλέπουμε 95 κράτη εδώ. Μας φαίνεται σημαντικό αριθμό. Θα πρέπει όμως να λάβει υπόψη το γεγονός ποιο είναι το σύνολο ή το ε, ποσοστό υιοθεσιών σε διεθνέ περίπτωση. Δεν θα αναφέρω τέτοιου είδου θέματα, αλλά πρέπει να πω ότι μειώθηκε ο αριθμό και στην πραγματικότητα περίπου 6% από τις υιοθεσίες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται στα πλαίσια της ε, Σύμβασης της Χάγης. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να πω ότι έχουμε 35 με 40% των υιοθεσιών που γίνονται εκτός, δεδομένου ότι γίνονται μεταξύ χωρών που δεν έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη. Αυτό όμως το ποσοστό σιγά σιγά αυξάνεται. Τα κράτη που δεν είναι μέρη της σύμβασης αυτής της στιγμής είναι η Ρωσία, η Αιθιοπία, η Κορέα και η Ουκρανία. Πήγαμε στην ε, Κορέα πριν από λίγο που πραγματικά υπέγραψε τη σύμβαση και περιμένουμε επικύρωση. Επίσης έχει επιδεικτεί ενδιαφέρον από την Ουκρανία και ελπίζουμε ότι το ποσοστό αυτό σιγά σιγά θα μειωθεί. Τώρα, ας έρθουμε στο τεχνικό θέμα το σημερινό. Τι σημαίνει αυτόματη αναγνώριση. Όπως ήδη προανέφερα, η αυτόματη αναγνώριση σημαίνει ότι έχουν γίνει σεβαστές οι εγγύησεις που προβλέπονται σύμφωνα με την ε, ε, σύμβαση. Δεν χρειάζεται λοιπόν η αναγνώριση, η εκτέλεση, η καταγραφή και για να διευκολυνθεί η κατάσταση υπάρχει ένα πιστοποιητικό πρότυπο το οποίο ακολουθούν οι χώρες που έχουν προσυπογράψει. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για πρώτα απ' όλα για τις υιοθεσίες. Δημιουργείται μία σχέση μεταξύ υιοθετούμενου και υιοθετηθέντος. Υπάρχει ε, μία ε, ευθύνη μεταξύ των ε, γονέων και ε, υπάρχει αυτό το οποίο λέγεται πλήρης υιοθεσία, νομίζω ότι είναι ε, σημαντικό να το αναφέρω. Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ αυτό που αναφέρουμε, απλή υιοθεσία ή πλήρης υιοθεσία και οι δύο καλύπτονται από τη σύμβαση κάθε φορά που υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετούμενη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι είδαμε στην αρχή του σεμιναρίου πως ε, πολλές χώρες σκέφτονται πόσο σημαντικό είναι να υποστηριχθούν οι βιολογικές οικογένειες. Όλο και περισσότερα ε, όλο και περισσότερο έχουμε ε, περιπτώσεις παιδιών που μεγαλώνουν και θα πρέπει να δούμε στο μέλλον κατά πόσον τέτοιου είδους ανοιχτές ιδιοθεσίες ε, στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα να έχει σχέση το παιδί με, τις, ε, με τη βιολογική του οικογένεια ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, ε, ενισχύσουμε. Επίσης, μιλήσαμε για μία αναγνώριση. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Η μία αναγνώριση είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει θέμα δημόσιας τάξης ή δεν προασπίζονται τα συμφέροντα του παιδιού. Η μία αναγνώριση της υιοθεσία είναι μία ε, ίστατη κύρωση για εξαιρετικές περιπτώσεις. Όταν ε, φερρυπίν υπάρχει απαγωγή του παιδιού, τότε δεν αναγνωρίζεται η υιοθεσία του. Επίσης, νομίζω ότι σε όλες τις ε, χώρες με τις οποίες ασχολούμαι. Εγώ έθεσα το ερώτημα εάν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μη αναγνωρισμένης υιοθεσίας και μου είπαν ότι λίγες. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Τι σημαίνει με τη σύμβαση αυτή. Έχουμε μία ενιαία διαδικασία μια πιο ταχεία διαδικασία, πιο απλή, λιγότερο δαπανηρή, μας δίνει την βεβαιότητα και την νομική ασφάλεια και όλα αυτά θεωρούνται από τα κράτη-μέλη σαν ε, θέματα τα οποία συνάδουν προς το να πούμε ότι πρόκειται για μια σύμβαση επιτυχή. Βεβαίως υπάρχουν και προβλήματα και αδυναμίες. Σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προσπάθειες σε κάθε χώρες ώστε να έχουμε καλύτερα πιστοποιητικά σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι αυτόματη η αναγνώριση εάν δεν υπάρξει εθνική αναγνώριση αθώμητα. Και αυτό είναι μία αδυναμία της συνθήκης της Χάγης και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Στην ε, περίπτωση παραβίασης ή προβλήματος που υπάρχουν με την υιοθεσία. Εμείς δεν νομίζω ότι έχουμε ένα δικαστήριο που μπορεί να εποπτεύει τέτοιου είδους καταστάσεις και να επιτηρεί τέτοιες καταστάσεις. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς σε περίπτωση όμως παραβίασης της όλης διαδικασίας είναι να έχουμε, όταν αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, να έχουμε συνεδριάσεις τρεις-τέσσερις φορές ε, ετησίως των κρατών που έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη και συζητούμε και μπορούμε να κάνουμε συστάσεις για το μέλλον, να μιλήσουμε για τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν και να προτείνουμε καινοτόμες λύσεις. Τρίτο μέρος, για να τελειώσω. Ποια είναι η περούσα κατάσταση. Έχουμε τις υιοθεσίες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση, δεδομένου ότι έχουμε όλο και περισσότερα κράτη που έχουν προσπαθήσει. Επίσης θα πρέπει να, έχουμε, ε, να παρέχουμε στις χώρες στις οποίες θέλουμε να γίνεται σωστά η υιοθεσία την ε, τεχνική υποστήριξη και έχουμε και άλλες διεθνείς υιοθεσίε που γίνονται εκτός σύμβασης Εκτός από τη Σύμβαση της Χάγης, αυτό που πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν προσπάθειες ώστε να προσχωρήσουν σε αυτή τη σύμβαση οι χώρες αυτές. Και αυτό μέσω τεχνικής βοήθειας που ήδη είναι ένα σύστημα το οποίο ακολουθήθηκε και δούλεψε στο παρελθόν. Επίσης, για πιο λεπτά και ευαίσθητα θέματα στις διάφορες ε, συνεδριάσεις που έχουμε θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι το 1993 ο κόσμος ήταν εντελώς διαφορετικός και οι απόψεις που υπερίσχυαν διαφορετικά. Σήμερα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, έχουν αλλάξει πολύ και θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η Σύμβαση της Χάγης είναι ένα, μια ζωντανή σύμβαση αν θέλετε η οποία πρέπει να εξελίσσεται αν συμφωνήσουν όλοι οι προσυπογράφοντες. Τι συμβαίνει τώρα με τις εθνικές υιοθεσίες που το εξετάζουμε σήμερα. Δεδομένου ότι βλέπουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε σε διεθνές επίπεδο και σήμερα τα έχουμε δεν υπάρχει αναγνώριση, αλλά θα ήθελα να καλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεωρήσει ότι το θέμα αυτό είναι ένα σφαιρικό πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει μόνο η Ευρώπη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες του κόσμου. Εάν έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα σφαιρικό, εάν θέλετε θα πρέπει να βρούμε και σφαιρική λύση. Διότι εάν κάνουμε κάτι για να ε, ρυθμίσουμε το πρόβλημα μόνο στην Ευρώπη, εξαιτίας των μεταναστευτικών ροών σε μερικά χρόνια το πρόβλημα αυτό θα ξαναπαρουσιαστεί στην Ευρώπη. Μία από τις προτάσεις μου είναι γιατί να μην κάνουν μία συνάντηση από κοινού τα κράτη-μέλη να προτείνουν το θέμα αυτό ως θέμα το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί από τα κράτη της Σύμβασης της Χάγης για να βρεθούν λύσεις λαμβάνοντας υπόψη τις, όλες τις ε, συμβάσεις από το 60, το 66 έως το 93 να δούμε ποια είναι τα ωφέλη που έχουμε αποκομίσει, ποια είναι τα θετικά στοιχεία, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποια είναι τα, είναι, είναι οι προκλήσεις και ποιες είναι οι λύσεις που πρέπει να υιοθετήσουμε για να ξεπεράσουμε αυτά τα θέματα προς συμφέρον των παιδιών. Πιστεύω ότι έχουμε την εμπειρία μας, την πρακτική, τους εμπειρογνώμονες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν και έχουμε για ένα θέμα το οποίο δεν είναι θέμα στο οποίο μπορούν πολλοί να ε, πουν κάτι αντίθετο, δεδομένου ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Νομίζω ότι έχουμε σε αυτά τα θέματα διεθνούς υιοθεσίες ε, πολλά, άρα θα πρέπει και σε εθνικό επίπεδο και για επιμέρους θέματα, όπως είναι αυτό των παρένθετων μητέρων Φερρυπίν, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση για να βοηθηθούμε όλοι περισσότερο. Ευχαριστώ. Ε, Σας Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρτίνες Μόρα. Θα σας παρακαλούσα να συγκεντρωθούν συζήτηση. Έχουμε καθυστέρηση 17 λεπτά που θα πρέπει να την καλύψουμε. Θα έλεγα να, πάρουμε, να πάρετε το λόγο μετά από τις παρεμβάσεις των κυρίων Ρωμάνο και Μόρα και μετά να συνεχίσουμε. Ερωτήσεις. Ο κύριος Γιάρα. Πολύ σύντομα μια ερώτηση αφορά ουσιαστικά τις ε, υιοθεσίε που γίνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη, τη συνένεση των γονέων. Αυτό φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει παραδείγματο χάρη σε διεθνέ επίπεδο, αλλά άκουσα αυτό που συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Το θεωρείτε καλό. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό γιατί έχουμε πολλές αναφορές στην Επιτροπή Αναφορών που αφορούν τέτοιες υιοθεσίε χωρίς συνένεση των γονέων. Ποια είναι η άποψή σας? Ευχαριστώ. Πράγματι είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Μία ερώτηση ακόμα. Επειδή σχεδόν όλες οι χώρες κύρωσαν τη σύμβαση του 1993, το δικό μας σημείο εκκίνησης δεν θα μπορούσε να είναι αυτή η συμφωνία με, αυτές, με τις διατάξεις της που είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι σημείο εκκίνησης για να υπάρξουν ευρωπαϊκές ε, διαδικασίες υιοθεσία. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς τον καθηγητή. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένας ενιαίος ορισμός, ορισμός ορισμένων θεμάτων που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο. Θα μπορούσατε ενδεχομένως να κάνετε κάποια πρόταση για μια σταδιακή διαδικασία, μια πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ό, το Συμβούλιο, έτσι ώστε να γίνει ενιαίο το δίκαιο σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το θέμα της υιοθεσία, θα ήθελα να πω ότι δεν θα πρέπει να συγχαίουμε μία διεθνή ε, υιοθεσία ε, με μία υιοθεσία που, από άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές ε, κουλτούρες. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που το θέμα είναι η διεθνή σύμβαση, σύμβαση δεν είναι υιοθεσία μέσα στη χώρα γιατί το παιδί βρίσκεται τη χώρα όπου υποβάλλεται το αίτημα υιοθεσία. Η κυρία Μαρτίνε θα μπορούσε να σα διαφωτίσει περαιτέρω τα πράγματα. Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Πρόεδρο σε ό,τι αφορά ορισμένε συστάσει που θα μπορούσα να κάνω. Δίχω άλλο θα ήταν πολύ δύσκολο να καταστήσει κανεί σε το Το δίκαιο. Βεβαίως η εναρμόνιση δεν μπορεί να αντικαταστήσει το εθνικό δίκτυο. Εδώ και μερικά χρόνια υπήρξε ένας κανονισμός ευρωπαϊκός που αφορούσε διεθνείς ε, ε, πωλήσει που δεν αντικατέστησε βεβαίως το εθνικό δίκαιο που κάλυπτε το θέμα των πωλήσεων ένα Γάλλο-Γερμανικό, Γάλλο-Λιθωνικό, Γάλλο-Πολωνικό, Γάλλο-Ισπανικό, ζευγάρι, Ισπανοϊρλανδικό ε, πολύ σύντομα θα έχει το δυνατότητα να συνάπτει έναν ευρωπαϊκό γάμο. Δηλαδή όσα να παντρεύεται ένας Γάλλος, μια Γαλλίδα, ένας Ισπανός, μια Ισπανίδα. Νομίζω ότι το μέλλον, στο μέλλον θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, ας παραμείνουμε στο παρόν. Νομίζω ότι με κάθε κόστος θα πρέπει να αποφύγουμε μία σύγκρουση των ε, δικαίων ότι δεν υπάρχει μία λύση. Δεν θα πρέπει να επανέλθουμε στον νόμο της ζούγκλας. Θα πρέπει να αποφύγουμε άτομα τα οποία ε, κινούνται στα πλαίσια μιας οικογενειακής σχέσης δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Πώς θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει βεβαίως να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα γιατί ήδη βρισκόμαστε πιο κοντά στη λύση. Αυτό που είναι ρεαλιστικό σήμερα είναι να επιτρέψουμε για λίγο καιρό ακόμα στις χώρες να είτε μιλάμε για ε, παρέθετη μητέρα είτε για μιλάμε, για, μιλάμε για γάμο ε, μεταξύ ατόμων του ιδίου φίλου να μπορούν να προχωρήσουν αλλά ο, το εφαρμοστέο δίκτυο σε αυτές τις περιπτώσεις για παράδειγμα υποχρέωση διατροφής ε, ε, ή θέματα κληρονομικά ο κανονισμός 650 του 2012 Εκεί θα πρέπει οι, οι, χώρες σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά να μην υπάρχουν συγκρουσιακές καταστάσεις ε, το... Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που όλα αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Εγώ ε, στρέφομαι προς τους νέους γιατί το μέλλον του ανήκει, η Ευρώπη του ανήκει. Αν πιστεύουν ότι σήμερα δεν είναι αποδεκτό στην Ευρώπη ένα διαζύγιο που έχει αποφασιστεί μεταξύ ενός Σουηδού και μίας Ιρλανδής δεν μπορεί να αναγνωριστεί στην Ιρλανδία. Δηλαδή το διαζύγιο να είναι ένα χολό διαζύγιο για την Ιρλανδία. Δηλαδή ο κύριος και η κυρία Τάδε να συνεχίζουν να είναι παντρεμένοι. Το να επιβάλλουμε μια μηδέα ε, αναγνώριση είναι κάτι απόλυτα εφικτό και θα είναι βεβαίως και αναγκαίο. Ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάσω το άρθρο 4 γάμα 1 που αφορά την συνένεση. Αναφέρεται ότι όλα τα άτομα, οι θεσμοί, οι αρχές, των οποίων απαιτείται η συνένεση για την υιοθεσία, την χάνουν της ε, σχετικής ενημέρωσης και βοήθειας όσον αφορά το τι σημαίνει η συνένεσή τους. Άρα, εδώ εξασφαλίζονται τα ελάχιστα ε, κατόφλια, αν θέλετε, εγγύσεων από τη της Το εθνικό δίκαιο είναι αυτό που θα αποφασίσει. Δηλαδή, Εάν συνενε... Δηλαδή, πρέπει να συνενέσει η βιολογική μητέρα. Δεν το λέει αυτό η Συνδίκη τη Χάγη, αλλά αυτό το οποίο λέει και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η βιολογική μητέρα πρέπει να έχει ενημερωθεί και να τύχει της ε, ειδική τεχνικής υποστήριξης και βοήθειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαφέρει από κάθε χώρα. Όταν όμως δίδεται η σωστή ενημέρωση, όταν ε, ενημερώνεται, συνοδεύεται ε, από κάποιον, όταν της πει κάποιος ποια είναι, ε, πώς μπορεί να βρει δουλειά, Φερρυπίν, όχι μόνο για ένα μήνα, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έχουμε την δυνατότητα να κρατήσει το παιδί της η μητέρα ή αν το δώσει προς υιοθεσία θα το δώσει αφού έχει ενημερωθεί και όχι μόνο διότι την πιέζει μια κατάσταση και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και θέλει χωρίς να το σκεφτεί δύο φορές να κάνει κάτι για να απαλλαγεί αυτή την κατάσταση πίεσης. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει υποστήριξη, βοήθεια και ενημέρωση. Αυτό ήθελα να τονίσω και πάλι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν να, περάσουμε στο επόμενο θέμα. Θα αναφερθούμε σε εθνικές υιοθεσίες και στην αναγνώρισή τους Χάρη στην κινητικότητα των ε, Ευρωπαίων πολιτών, παραδείγματο χάρη να μετακομίζει μια οικογένεια που έχει υιοθετήσει ένα παιδί. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην κυρία Καμπέζα. Είναι μέλος ενός ε, διεθνούς οργανισμού νομικών συμβούλων. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ για να μιλήσω για αυτό το θέμα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Και θα ξεκινήσω με τα πρώτα απορίσματά μου. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να ξεκινήσω από αυτό είναι ότι δεν υπάρχει σήμερα μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει τη δυνατότητα είτε να υπάρξει αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση είτε εκτέλεση κάποιων αποφάσεων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, γιατί άκουσα τον πρώτο μιλητή, ο οποίος ανέφερε το θέμα της μη ύπαρξης ενός επιπλέον συμβατικού κειμένου, καθότι έχουμε τη σύμβαση της ΧΑΗΣ του 1993 και λέει ότι ουσιαστικά οι υιοθεσίε ε, διακρατικές στην ευρύτερη έννοια δεν δημιουργούν προβλήματα καθότι υπάρχει αυτή η σύμβαση του 1993. Όμως ε, τελικά από ό,τι είδαμε από τις παρουσιάσεις κάποιων άλλων ομιλητών τι σημαίνει ακριβώς αυτή η διακρατική υιοθεσία. Και όπως ξέρουμε Εκεί προκύπτουν τα προβλήματα, όπως παραδείγματο χάρη η οικογένεια που υιοθετεί βρίσκεται σε μία χώρα και το παιδί ζει σε μία άλλη χώρα. Ο τόπος διαμονής παραδείγματο χάρη ε, έχει σχέση με τον ορισμό αυτό και όχι η ηθαγένεια. Σύμφωνα με το Βρετανικό δίκαιο, με το Αγγλικό δίκαιο, μία υιοθεσία στο εσωτερικό μιας χώρας δεν εξαρτάται ούτε από τον τόπο διαμονής, ούτε από την ηθαγένεια, ούτε από το που διαμένει η οικογένεια που θέλει να υιοθετήσει. Είναι λοιπόν δυνατόν, σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο, να πάρει την απόφαση για μια υιοθεσία για ένα παιδί που ζει σε μια άλλη χώρα και να γίνει η υιοθεσία από οικογένεια, από γονείς, που ζουν στην ίδια χώρα με το παιδί προς υιοθεσία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος ζει στην Αγγλία, προσωρινά όμως διαμένει στη Γαλλία, με έναν Γάλλο αποφασίζει να υιοθετήσει ένα παιδί στη Γαλλία. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί η απόφαση να ληφθεί από ένα αγγλικό δικαστήριο. Έχει λοιπόν αρμοδιότητα το Βρετανικό δικαστήριο για ένα παιδί που ζει στη Γαλλία από τη στιγμή που ένας από τους δύο γονείς είναι Βρετανός υπήκος. Αυτή η απόφαση φυσικά είναι με το αγγλικό δίκαιο όμως δεν αναγνωρίζεται αυτόματα από τις γαλλικές αρχές. Άρα, αυτό που σκεφτόμουν, και αυτό είναι και οι ιδέες που παρουσιάζω στο έγγραφό μου, είναι ότι αν πρέπει να υπάρξει κάποια αναγνώριση, κάποια ρύθμιση, αν πρέπει λοιπόν να υπάρξει αναγνώριση, πώς αυτό θα πρέπει να γίνει. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η αναγνώριση θα πρέπει να γίνεται με αυτόματο τρόπο είτε με συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν θα διαβάσω όλο μου το έγγραφο, αλλά αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Υιοθεσία των Παιδιών, τα ελάχιστα προαπαιτούμενα και τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει, 10 ευρωπαϊκές χώρες. Ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε στις ε, περιπτώσεις αυτές που δεν αναγνωρίζονται οι αποφάσεις των ε, ξένων δικαστηρίων, Αναφέρεται επίσης η γονική ευθύνη, θέματα φορολογικά, το που διαμονείς. Όλοι αυτοί οι λόγοι μπορεί να οδηγήσουν στη μη αναγνώριση και υπάρχει σαφής ασάφεια στο κανονισμό Βρυξέλλες 2Β. Καθότι το θέμα της υιοθεσία και της γονικής ευθύνης σε περιπτώσεις που μια χώρα, παραδείγματο χάρη, δεν αναγνωρίζει μια απόφαση για υιοθεσία, δεν μπορεί βεβαίως κατ' επέκταση και να αναγνωρίσει τη γονική ευθύνη. Χωρίς την απόφαση της υιοθεσία δεν υπάρχει γονική ευθύνη. Στο έγγραφό μου, λοιπόν, χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα τεχνητό και αναφέρομαι σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς να θέλω να αναφερθώ ρητά σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά αν κάποιος θέλει να υιοθετήσει ένα παιδί και ζει στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, σε μια άλλη χώρα με το παιδί του, το θέμα είναι αν μπορεί, λόγω της μη αναγνώρισης, παραδείγματο χάρη, να ε, προσφέρει στο παιδί του ιατρική περίθαλψη. Όπως ξέρετε, από τη στιγμή, παραδείγματο χάρη που προχωρήσει η οθεσία, το παιδί παίρνει ένα διαβατήριο με το όνομα των γονέων. Σε αυτή την περίπτωση δεν ε, προκύπτει θέμα αν πρόκειται για υιοθετημένο παιδί ή φυσικό παιδί. Μπορεί όμως να προκύψει εάν ένας από τους δύο γονείς δεν έχει γονική ευθύνη, είτε εάν παραδείγματο χάρη πρόκειται για δύο γονείς του ίδιου φίλου ή εάν υπάρχει ε, διαφορετική ε, προέλευση οι γονείς και το παιδί προέρχονται από διαφορετική χώρα. Προτείνω λοιπόν και κάποιες λύσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι δυσκολίες, ποια είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Είναι τα βασικά ερωτήματα που θα ήθελα να σας αναφέρω για να τα σκεφτείτε. Εάν υπάρχει αυτόματη αναγνώριση από όλα τα κράτη-μέλη, κάποιων αποφάσεων που λαμβάνονται από ένα εθνικό δικαστήριο, αυτή είναι, αν θέλετε, η πιο ριζοσπαστική λύση. Αυτό με την αναγνώριση από όλε τι χώρε. Και αυτό βεβαίω σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολα αποδεχτή, καθότι υπάρχουν χώρες, παραδείγματος χάρη, που δεν δέχονται την υιοθεσία παιδιού από ένα ζευγάρι του ίδιου φίλου. Μια άλλη εναλλακτική που προτείνω είναι λιγότερη, αν θέλετε, λιγότερο ριζοσπαστική. Ένα δικαστήριο παίρνει μια απόφαση και θα πρέπει να αναγνωρίζετε αυτόματα από την χώρα στην οποία το παιδί έχει τον συνήθι τόπο διαμονής του. Βάσει βεβαίως αυτόν που ορίζει η σύμβαση της Χάγης του 1993, καθότι η απόφαση αυτή έχει σαν σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Άρα ο τόπος διαμονής ε, του παιδιού προς υιοθεσία που αποτελεί ένα από τα κριτήρια της Σύμβασης της Χάγης Ο τόπος συνήθως διαμονής λοιπόν του παιδιού και σε περίπτωση που η απόφαση ληφθεί από ένα δικαστήριο μιας άλλης χώρας καθότι ένας από τους δύο άλλους γονείς είναι υπήκος μιας άλλης χώρας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει αυτόματη αναγνώριση του κράτους μέλους συνήθως ε, τόπου διαμονής της χώρας. Τώρα, αν το παιδί έχει διαφορετική ηθαγένεια από αυτήν του τόπου διαμονής του. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως θα πρέπει η απόφαση οθεσίας να αναγνωρίζεται μόνο από την χώρα του συνήθους τόπου διαμονής του παιδιού. Και σε κάθε περίπτωση, εάν και εφόσον το κράτος μέλος διαμονής δεν είναι το κράτος μέλος διαμονής των γονέων. Το παράδειγμα που σας έδωσα προηγουμένως, ένα παιδί το οποίο διαμένει στη Γαλλία με μια μητέρα, της οποίας ο συνήθως τόπος διαμονής είναι η Μεγάλη Βρετανία και σε αυτή την περίπτωση το δικαστήριο το Βρετανικό παίρνει μια απόφαση η οποία θα πρέπει να αναγνωριστεί και να γίνει δεκτή και από την Γαλλία αυτόματη λοιπόν αναγνώριση μιας απόφασης και σε περίπτωση ηθαγένειας, διαφορετικής ηθαγένειας ενός παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προβλέπετε μια διαδικασία, αν υπάρχει δικαστική συνεργασία μεταξύ των αρχών και βεβαίως βάσει των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που θέτει η Σύμβαση της ΧΑΗΣ το 1993 και εδώ βεβαίω δεν πρόκειται για διακρατικές υιοθεσίε, αλλά για υιοθεσίε στο εσωτερικό μια χώρας. Νομίζω ότι όλε αυτέ οι δυσκολίε θα πρέπει να ξεπεραστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια χώρα που απαγορεύει, παραδείγματο χάρη την υιοθεσία από ζευγάρια του ίδιου φίλου, θα υιοθετήσει μια διαδικασία υιοθεσία τέτοιου τύπου που λαμβάνει η χώρα σε μια άλλη σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό θα είναι βεβαίως ένα μειονέκτημα όσον αφορά την, ε, τον αριθμό των υιοθεσιών που θα αναγνωρίζονται. Απ' την άλλη για το ίδιο το παιδί αυτό μπορεί να είναι κάτι το θετικό καθότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση βάσει της σύμβασης του 1993 για τις υιοθεσίε στο εσωτερικό μιας χώρας θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του παραδείγματος χάνει για μια υιοθεσία στην Αγγλία και αφορά ένα παιδί που ε, διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία, αλλά είναι, έχει την πολωνική ηθαγένεια. Σε κάθε περίπτωση οι πολωνικές αρχές θα πρέπει να ενημερώνονται όσον αφορά την υιοθεσία, τις ε, προϋποθέσεις και να τους δίνεται η δυνατότητα να συνεισφέρουν, να συμμετέχουν στη διαδικασία της υιοθεσία στην Μεγάλη Βρετανία. Αλλά ο Βρετανός δικαστής δεν ε, θα πρέπει να δεσμεύεται από την απόφαση των πολωνικών αρχών σε αυτή την περίπτωση. Το 1996, στο άρθρο 33, αναφέρεται η υποχρέωση διαβούλευσης με την ε, άλλη χώρα. Παραδείγματος χάρη η απόφαση του Βρετανικού Δικαστηρίου για ένα μέλος μιας οικογένειας που ζει στην Αυστραλία, για ένα παιδί που ζει στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερωθεί, να υπάρξει διαβούλευση και το μέλος οικογένειας που ζει στην Αυστραλία υποχρεούται να δεχθεί την απόφαση. Υπάρχει λοιπόν διαβούλευση, ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά όχι υποχρέωση δεσμεστική όπως ε, ορίζει το άρθρο 17 της Σύμβασης του 1993. Και αυτός είναι ένας άλλος τρόπος ενδεχομένως να αντιμετωπίσει κανείς την ε, αναγνώριση. Τέλος, η αυτόματη αναγνώριση σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το απαιτήσουμε δεδομένης της μεγάλης αν θέλετε, διαφοράς που συνεχίζει να υπάρχει στα νομικά συστήματα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία για αναγνώριση. Σήμερα διαφορετική νομοθεσία διέπει την διαδικασία αναγνώρισης. Ενδεχομένως θα μπορούσε αυτό να εναρμονιστεί. Να υπάρχει μία ενιαία διαδικασία για την αίτηση για την αίτηση αναγνώρισης και να υπάρχει μία απόφαση ναι ή όχι όσον αφορά το αποτέλεσμα. Αλλά τουλάχιστον οι γονείς θα είναι σαφείς όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν και θα έχουν μία απόφαση ναι ή όχι και δεν θα έχουν άχρηστες διαδικασίες, ατέρμονες και δαπανηρές Εξάλλου η πραγματικότητα, ιδιαίτερα για παιδιά τα οποία ζουν σε μια άλλη χώρα, και σήμερα γνωρίζουμε ότι οι οικογένειες στην Ευρώπη μετακομίζουν, αλλάζουν τόπο διανομής για οικογενειακούς λόγους, για <laughs> επαγγελματικούς λόγους. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει νομική ασφάλεια, να υπάρχει βεβαιότητα όσον αφορά την αρμοδιότητα για τις αποφάσεις. Ποιος είναι αρμόδιος. Ιδιαίτερα για οικογένειες που μετακομίζουν και ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καμπέζα. Πραγματικά θαυμάσια η παρέμβασή σας στη συζήτησή μας. Αυτό είναι ένα θέμα που περιπλέκεται όλο και περισσότερο στο μυαλό μου μετά από τις διάφορες παρεμβάσεις που ακούστηκαν. Όλο και μεγαλύτερη τρικυμία στο κρανίο μου. Αλλά θα πρέπει να μην ξεφεύγουμε από τον βασικό μας στόχο, το συμφέρον του παιδιού. Ενδεχομένως τα νομικά προβλήματα θα μπορούσαμε να τα λύσουμε με μεγαλύτερη ευκολία. Από την άλλη βεβαίως Γνωρίζουμε ότι υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό, η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μόνο και έχουμε πάντοτε προβλήματα με αυτή την ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όταν δούλευα το Βρυξέλλες 1 Κάναμε αναφορά στην αναγνώριση των αποφάσεων στα πλαίσια του αστικού ή του εμπορικού δικαίου και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς ε, τις άλλες νομοθεσίες των άλλων χωρών. Είναι λοιπόν ένα πραγματικό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση θα το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Έχουμε έναν άλλο εμπειρογνώμονα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι μιλάμε για προβλήματα υιοθεσία στην Ευρώπη, ξεχνώντας ότι υπάρχουν χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει ο θεσμός της υιοθεσία. Η κυρία Νάτσμα Γιασάρη, που εργάζεται στο Ινστιτούτο Max Planck, θα μας ε, μιλήσει για τη Μέση Ανατολή και τα μέσα που υπάρχουν για την προστασία των ανηλίκων. Δεν αφορούν υιοθεσίε αυτά τα μέσα, αλλά ε, προστασία κυρίως. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψε μου να σας οδηγήσω μακριά από την Ευρώπη. Στόχος μας είναι να δούμε την υιοθεσία, αλλά κανένας από εμά δεν όρισε την υιοθεσία. Χρησιμοποιούμε χιλιάδες χρόνια τον όρο υιοθεσία και το περιεχόμενο της υιοθεσία έχει αλλάξει και έχει εξελιχθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε το θέμα αυτό για να καταλάβουμε την ουσία των νομικών πτυχών που θέλουμε να κατανοήσουμε ή να μεταγράψουμε. Και αυτό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα διαφορετικά νοήματα. Έχουμε λοιπόν προβλήματα στην αναγνώριση της υιοθεσία, ό,τι και να σημαίνει. Από την Ιταλία στη Γαλλία, από την Γαλλία στην Ιταλία ε, και πολλά άλλα. Ε, εγώ σπούδασα νομικά στην Αυστρία και στην Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία εξετάζοντας τους ορισμούς που θα βρείτε θα έλεγα ότι δεν θα έπρεπε να γνωρίζετε μια αυστριακή υιοθεσία γιατί είναι εντελώς διαφορετική από τον τρόπο που γίνεται αντιληπτή στη Γερμανία. Ακούσαμε ότι είναι μια αντιστρέψιμες υιοθεσίες. Υπάρχει η ανάκληση, προβλέπεται η ανάκληση της υιοθεσίας στη Γερμανία, στην Αυστρία, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπάρχει η επιλογή της ανάκλησης. Το θέμα λοιπόν είναι τι είναι η υιοθεσία. Ε, εγώ ασχολήθηκα με την έρευνα και θα ήθελα να τα αναφέρω αυτά και να πω πόσο σημαντικό είναι το συγκριτικό δίκαιο για να μπορέσουμε να δούμε το πώς η κάθε χώρα κατανοεί το θέμα της υιοθεσία. Μετά από την έρευνά μου κατέληξα σε ορισμένα βασικά στοιχεία της υιοθεσία που έχουν τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι σε σχέση με την ιστορική εξέλιξη της υιοθεσία, σήμερα η υιοθεσία πρωτίστως δεν αφορά τη μεταφορά του οικογενειακού ονόματος ή της οικογενειακής περιουσίας και δεν γίνεται πρωτίστως μεταξύ ενηλίκων όπως γινόταν ιστορικά. Σήμερα η υιοθεσία στόχο έχει να δημιουργήσει ένα καινούριο νομικό δεσμό μεταξύ των γονιών και του παιδιού σε μόνιμη βάση και με τον όρο μόνιμος εννοούμε ότι αυτό ο δεσμός δεν τελειώνει με την ελικίωση του παιδιού έχει στόχο να δώσει ε, ε, γονική κυριαρχία ή μέρημνα και στους δύο γονείς ή μάλλον κυριαρχία ε, και όρος αυτός περιλαμβάνει ε, πάρα πολλά όλα τα, περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα, όλες τις υποχρεώσεις που έχει ένας βιολογικός γονιός προς το βιολογικό του παιδί. Αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η ευημερία του παιδιού. Είναι δυνατός λοιπόν, είναι διαιτή μόνο μόνον αν είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Εκεί δεν ορίζεται ε, λεπτομερώς ε, η υιοθεσία, απλά και μόνο αναφέρεται ότι πρέπει να είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Εάν λοιπόν καταλήξουμε ότι μιλάμε μιλώντας για την υιοθεσία μπορεί ο καθένας μας να εννοεί διαφορετικά πράγματα θα πρέπει να βρούμε ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Η επικοινωνία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να επικοινωνούμε με τις ίδιες λέξεις αλλά να εννοούμε διαφορετικά πράγματα. Και εκεί χάνεται η επικοινωνία. Αν λοιπόν να συμφωνήσουμε ως προς τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορείτε βεβαίως να αφισβητήσετε, θα μπορούσαμε να περάσουμε σε νομικές ε, ε, δομές που υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Εμένα με απασχολούν οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά αυτές αυτές τις χώρες και θα σας εκπλήξουν αυτά που έχω να σας πω. Θα ξεκινήσω με κάτι που βρίσκεται στο κέντρο της έρευνάς μου και αυτό είναι κάτι που θέλω να το δημοσιοποιήσω. Το καφάλα είναι ένας όρος του Ισλαμικού δικαίου και εγγυάται έναν δεσμό. Το υιοθέτησαν οι χώρες της Βόρειας Αφρικής, κυρίως η Τινησία το Μαρόκο και η Αλγερία βρίσκεται και στο Σουροζάν και στην Αίγυπτο. Δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ε, μουσουλμανικό δίκαιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η ιδέα ότι υπάρχει καφάλα και δεν υπάρχει οθεσία είναι λάθος. Αυτό είναι ε, ένα σημαντικό σημείο. Δεύτερον, Καφάλα δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα και στις τρεις χώρες που ανέφερε την Ισία, Αλγερία και Μαρόκο. Γιατί, όπως σας είπα, είναι πολύ σημαντικέ οι λεπτομέρειε, Για την Ισία, με και στο Μαρόκο, το καφάλα τελειώνει με την ενηλικίωση του παιδιού. Θα μπορούσε, ας πούμε, να θεωρηθεί κάτι παρόμοιο με το να είναι κανεί ανάδοχο ε, γονέας. Στην Αλγερία όμως δεν συμβαίνει. Βασίζεται στην ιδέα δημιουργίας μιας μόνιμης σχέσης. Επίσης, είναι σημαντική η έννοια τις ε, ε, θα πρέπει να πούμε ότι το γερμανικό δίκαιο χωριζόταν σε δύο μέρη. Το ένα αφορούσε τη φροντίδα ενός παιδιού, την ανατροφή και το άλλο αφορούσε τα περιουσιακά του στοιχεία. Και τα δύο αυτά μαζί αφορούν την γονική μέρημνα. Στην καφάλα όλο αυτό μεταφέρεται στο άτομο που αναλαμβάνει την καφάλα. Έχουμε λοιπόν δύο σημαντικά σημεία εδώ. Στον ορισμό ή στο αντίστοιχο ε, της ε, ε, ε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής διαπιστώσαμε ότι έχει έχουν ενσωματωθεί τα τελευταία 30 χρόνια η αρχή του συμφέροντος του παιδιού που είναι η πρωταρχική αρχή. Υπάρχουν και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στις χώρες αυτές υπάρχει το εθνικό δίκαιο και δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε στο προφήτη του, στο χατζή του, σε κανένα. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό γιατί υπάρχουν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το δίκαιο σε αυτές τις χώρες. Το πρόβλημα που έχουμε στην Αλγερία και υπάρχει ένας τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι ότι ο κώδικας στην Αλγερία αναφέρει η, ε, απαγορεύεται η οθεσία, Έτσι λέει ε, μεταφρασμένο. Ε, βεβαίως ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι το καμπάλι απαγορεύει, να χρησιμοποιείται η λέξη καμπάλι, δηλαδή οποιαδήποτε σχέση μεταφέρει όσα προκύπτουν από την υπαγωγή, απαγορεύεται σε αυτό το δίκαιο, δεν σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η οθεσία στην Αλγερία. Δεν λέω ότι ξέρω καλύτερα το πώς έχουν τα πράγματα από τον Αλγερινό νομοθέτη. Λέω όμως για ότι για λόγους ε, εσωτερικού δίκαιου στην Αλγερία εστιάζεται διαφορετικά τα πράγματα από ότι αν επρόκειτο για ένα ξένο. Χρειάζεται να το δούμε το πράγμα συγκριτικά για να καταλάβουμε. Αν το κάνουμε αυτό αυτό θα καταλήξουμε στο αποτέλεσμα ότι ως ε, δυτικός ε, δικαστής θα μπορέσει κανείς να αναγνωρίσει το καμπάλα ως απλή υιοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα όταν έχουμε να κάνουμε γενικά με θέματα που αφορούν την λειτουργία αυτής, ε, αυτού του θεσμού και σε τι χρησιμεύει και γιατί ο νομοθέτης ε, ενέργησε έτσι και πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό σε ένα διεθνές ε, πλαίσιο. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα είναι ο νόμος στο Ιράκ. Στο Ιρακινό δίκαιο έχουμε ένα νόμο νεανικής πρόνοιας που επιτρέπει τη μεταβίβαση του ονόματος στο παιδί και την μεταβίβαση ενός μέρους της ε, υιοθεσίας, της περιουσίας. Δηλαδή εδώ μιλάμε για πλήρη υιοθεσία. Είναι το ίδιο πράγμα σαν να επρόκειτο για μια βιολογική σχέση. Παρόλα αυτά, αν εξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο τα δυτικά δικαστήρια αντιμετώπισαν οποιονδήποτε προέρχεται από τη Μέση Ανατολή αντιμετώπισαν ε, ε, στα πλαίσια του Ισλαμικού δικαίου χωρίς να σκεφτούν το εθνικό δίκαιο και θεωρούν ότι οι χώρες αυτές είναι ένα ολόκληρο μπλόκο. Υπάρχουν χώρες που απαγορεύουν το καμπάνι, την ε, υιοθεσία, αλλά ε, δεν ε, παρέχουν κάτι αντίστοιχο. Αλλά αυτό αφορά αυτές τις χώρες. Ως ε, επειδή το συγκριτικό δίκαιο ε, είναι ο τομέας που με ενδιαφέρει, θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει η οθεσία για μας και για τους άλλους. Θα πρέπει λοιπόν να μεταφέρουμε την προσοχή μας από τις ταμπέλες στα πραγματικά γεγονότα. Όταν βρίσκουμε μια περίπτωση όπου το παιδί μπορεί να ενσωματωθεί σε μια οικογένεια μονίμως, ε, όπου να υπάρχει πλήρης γονική μπνε, μέρημνα υπάρχει η δυνατότητα να αναζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας υιοθεσία και αυτό στα πλαίσια του συμφέροντος του παιδιού. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε την ιδέα της προστασίας του παιδιού. Ε, ε, θα πρέπει πολύ συχνά το γερμανικό κράτος ε, ε, φέρει μια άποψη για την αναγνώριση της υιοθεσία χρησιμοποιώντας την ίδια, τον ίδιο ακριβώς τύπο. Λέει ας πούμε ότι το Κοράνι δεν αφήνει περιθώριο για την υιοθεσία. Θα μπορούσα να σας πω ότι στο Κοράνι δεν υπάρχει καμία αναφορά στην υιοθεσία. Η μόνη αναφορά είναι ότι ένα παιδί θα πρέπει να κρατάει την ταυτότητά του, θα πρέπει να φέρει το όνομα ε, του πατέρα του. Το δεύτερο σημείο αναφέρεται ότι ε, ε, τα εμπόδια για το γάμο που οφείλονται στη βιολογική ε, σχέση, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ στενών ε, συγγενών, ισχύει και στην περίπτωση της ε, υιοθεσία. Αυτό που απαγορευόταν τον, και το στο Ισλάμ ήταν διαφορετικό. Τότε την υιοθεσία γινόταν μεταξύ ενηλίκων που ανήκαν σε διαφορετικές φυλές. Ε, συνήθως η υιοθεσία γινόταν για να ε, μπορέσουν να, να, μπορέσουν να μεταφερθούν τα περιουσιακά ε, στοιχεία, η εξουσία ή εξουσία. Αυτό λοιπόν που εννοούμε σήμερα με τον όρο υιοθεσία δεν απαγορεύεται από το Ισλάμ. Είναι λάθος το να λέμε ότι το Κοράνι ε, απαγορεύει την υιοθεσία. Ε, ε, υπάρχει μια γενικότερη εντύπωση ότι ε, αυτό συμβαίνει, αλλά δεν είναι σωστό. Τώρα, αν συγκρίνουμε κάτι άλλο θα μπορούσαμε να παρεξετάσουμε την ε, ορολογία που χρησιμοποιείται και ενδεχομένως θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική διατύπωση, να προσθεθεί κάτι, να δώσουμε μια περιγραφή ε, της ε, Όχι να χρησιμοποιήσουμε απλά και μόνο τον όρο υιοθεσία. Το τελευταίο σημείο, γιατί και αυτό το θέμα ετέθη το, η σύμφωνη γνώμη των βιολογικών γονιών. Εδώ έχουμε ένα δίλημα. Μιλάμε για χώρες που επισήμως απαγορεύουν την υιοθεσία ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε χώρες ε, που ε, ε, απαγορεύουν την πλήρη υιοθεσία αλλά έχουν κάτι αντίστοιχο. Στο γερμανικό δίκαιο θα μπορούσε να υπάρχει υιοθεσία νόσηρα κοινού να, και να θεωρήσουμε ότι έγινε στο Ιράκ ε, και το παιδί είναι από το Ιράκ. Ε, το παιδί ε, μεταφέρεται στη Γερμανία και υποβάλλεται αίτημα για υιοθεσία. Το δικαστήριο λέει αυτή είναι μία δύναμη υιοθεσία. μία μερική υιοθεσία. Οι γονεί θέλουν να γίνει πλήρης η υιοθεσία αυτή. Ή μία χολή υιοθεσία. Θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτή την περίπτωση. Ε, αν πάρουμε το αντίστοιχο σε μια μουσουλμανική χώρα, μια υιοθεσία δηλαδή που δεν, είναι και που δεν επιτρέπει την πλήρη υιοθεσία και το μεταφέρουμε σε ε, πλήρη υιοθεσία, αλλά γι' αυτό χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της βιολογικής μητέρας, τι σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή θα πρέπει να συμφωνήσει με κάτι που απαγορεύεται στη χώρα σας. Θα πρέπει να πάει στην γερμανική πρεσβεία, στη Σταμπούλ και να πει ότι συμφωνεί να υπάρξει πλήρης υιοθεσία. Η γερμανική πρεσβεία στη Σαμπούλ μπορούν να πούν δεν μπορούμε να διδαχτούμε κάτι που είναι παράνομο στη χώρα σου. Ακόμα και αν θέλει λοιπόν να συμφωνήσει δεν μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε την ιδέα της αναγνώρισης που έχουμε και πώς ε, αντιμετωπίζουμε τις χώρες που δεν επιτρέπουν την πλήρη υιοθεσία. Εγώ δεν έχω καταλήξει σε κάποια λύση γιατί εδώ τίθεται αυτό το θέμα της ε, σύμφωνη γνώμη τη γυναίκα. Το Ισλαμικό δίκτυο, λοιπόν, ε, δίκαιο δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν εφαρμόζεται σε όλες τις μουσουλμανικές χώρε με εξαίρεση το οικογενειακό δίκτυο, δίκαιο που είναι η βάση του κωδικοποιημένου εθνικού δικαίου. Και νομίζω ότι κάθε φορά θα πρέπει να εξετάζουμε τη συγκεκριμένη χώρα της Μέσης Ανατολής. Θα μπορούμε ε, να είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι αφορά τον ορισμό της υιοθεσία. Αυτό που θέλουμε είναι μια στενή σχέση, τη μέρημνα του γονιού και το συμφέρον του παιδιού. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście niezwykle e, interesujący. Ναι, πρόκειται για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Βλέπετε τα πράγματα με μια διαφορετική, αν θέλετε, οπτική γωνιά. Ξεχνάμε ότι άλλα συστήματα μπορεί να μας επιτρέψουν ε, μια άλλη προσέγγιση. Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, έχετε το λόγο. Όχι, δεν βλέπω κανέναν να ζητάει το λόγο. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι φαίνεται. Χάρη σε όλες τις πληροφορίες που πήραμε. Νομίζω ότι η προσεγγίσεις μας διαφέρουν και θεωρώ ότι η νομοθετική εργασία που θα ακολουθήσει θα λάβει υπόψη πολλά από τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε σήμερα. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι το καλό του παιδιού είναι ο σκοπός όλων αυτών των προσπαθειών μας. Τώρα, όσον αφορά την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών ή μεταξύ διεθνών οργανισμών, τελικά όλα αυτά έχουν δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με την προστασία του παιδιού. Βέβαια θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση, να μειώσουμε τις διαφορές που βασίζονται πολλές φορές και οφείλονται στην παράδοση, στην ιστορία, στη θρησκεία και στη γλώσσα. Ας μην ξεχνάμε τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ του ορισμού της οικογένειας από τη μία χώρα στην άλλη παραδείγματος χάρη υιοθεσία από ζευγάρια του ίδιου φίλου, κάτι που δεν αναγνωρίζεται από πολλές χώρες. Υπάρχουν και τα θέματα υιοθεσία παιδιών από γονείς οι οποίοι βρίσκονται στη ζωή, είτε από γονείς οι οποίοι έχουν πεθάνει. Όλες αυτές οι πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη και πιστεύω ότι του χρόνου θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Βρυξέλλες 2α σίγουρα θα μας υποβληθεί πολύ σύντομα. Σήμερα εξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξ ονόματος όλων των συναδέλφων, μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ στις Βρυξέλλες για να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας. Είμαστε ευγνώμονες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία και ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση.